Hello everyone, good afternoon. Καλό απόγευμα σε όλους. Όσον αφορά την ημερήσια διάταξη, υπό το 4 θα προσθεθεί ένα νέο, ημερήσι, ένα νέο σημείο στην ημερήσια διάταξη, ε, έτσι ώστε να υπάρξει ενημέρωση για τις ε, διαπραγματεύσεις. Εάν συμφωνείτε με αυτή την τροποποίηση, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Έχω και κάποιες ανακοινώσεις. Στη συνάντηση της 5ης 21ης Φεβρουαρίου το απόγευμα, ε, αυτή δεν θα λάβει χώρα. Ε, οι συνεδριάσεις θα γίνουν 20 Φεβρουαρίου το πρωί και το, το απόγευμα και την 5η 21 Φεβρουαρίου μόνο το πρωί όπως ε, ε, έχουμε συμφωνήσει. Επίσης αλλαγές στην γραμματεία. Μετά από 10 χρόνια στη γραμματεία της ΕΝΒ η Εμίλια Ρωμάνο θα την εγκαταλείψει γιατί από την 1η Φεβρουαρίου θα γίνει επικεφαλής μονάδος στην υποστήριξη των Ιταλών ε, βουλευτών στην DGI Tech. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, να σας ενημερώσω επίσης ότι έχουμε 21 γλώσσες όσον αφορά το καθεστώς διερμηνίας. Επίσης ότι οι φάκελοι βρίσκονται διαδικτυακά διαθέσιμοι και επίσης ότι ε, η συνεδρίαση θα καταγράφεται στο διαδίκτυο. αυτές ήταν οι ανακοινώσεις. Να σας πω επίσης ε, τι έγινε με, τους, ε, με τα πρακτικά της συνεδριάσεως των συντονιστών. Ωραία. Ε, και αυτό εγκρίθηκε. Να σας πω τώρα δύο λόγια όσον αφορά τις διοργανικές διαπραγματεύσεις. Είχαμε δεύτερο τριμερή διάλογο την 22 η Ιανουαρίου ε, όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος για τα βαρέα οχήματα. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είχαν λεπτομερή συζήτηση όσον αφορά τις τροπολογίες που από τις δύο πλευρές είχαν κατατεθεί. Επίσης ε, ε, επιτύχαμε συμβιβασμό όσον αφορά τα λιγότερο πολιτικά ζητήματα όπως τα υποστηρικτικά μέτρα κτλ. Ε, το monitoring, την περίοδο επιθεώρησης και αναφοράς, την ανάλυση του κύκλου ζωής ε, κτλ. Ε, κάποια άλλα ζητήματα όπως, όπως είναι το EMS, όπως είναι εναλλακτικά καύσιμα, όπως είναι κάποιες κυβερνητικές διατάξεις και πολιτικώς ευαίσθητα θέματα και κυρίως τα κίνητρα για τα οχήματα μηδενικής ή χαμηλή, μηδενικών χαμηλών εκπομπών ε, θα γίνουν περαιτέρω συζητήσει. Όσον αφορά τώρα τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα ε, στην, ε, στην ανάλυση, αξιολόγηση κινδύνου στην διατροφική αλυσίδα τη Ευρωπαϊκής Ένωση. είχαμε το δεύτερο άτομο υποτριμερή διάλογο την Πέμπτη, την προηγούμενη εβδομάδα 24 Ιανουαρίου. Στο τριμερή διάλογο αυτό το Κοινοβούλιο προώθησε μία δέσμη προτάσεων σε σχέση με αρκετά πολιτικά ζητήματα σε μια προσπάθεια να αφήσει μόνο σε εκκρεμότητα ε, μερικά πολιτικής φύσεως ζητήματα για τον τρίτο τριμερή διάλογο. Το Συμβούλιο ε, αντιστρόφως έδειξε κάποια ευελιξία όσον αφορά τα εργαλεία για την επικοινωνία του κινδύνου, όσον αφορά επίσης τη σύνθεση ε, του Management Board της ΕΦΣΑ και όσον αφορά επίσης ε, την ε, συμπερίληψη ενεργών επιστημόνων στα πάνελ των επιστημόνων. Όσον αφορά τα καθαρά οχήματα, στον τριμερή διάλογο υποβάλαμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συμφωνήθηκε ότι τα κύρια πολιτικά ζητήματα ε, θα ε, ε, βρεθούν εντός του εύρους της οδηγίας. Ε, επίσης ε, θα γίνει και γίνεται λόγος επίσης και για τα καθαρά οχήματα καθώς επίσης ε, και για την περίοδο μεταφοράς. Επίσης συμφωνήθηκε ότι τα πολιτικά ζητήματα θα συζητηθούν σε τεχνικό επίπεδο έτσι ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος για περαιτέρω συζητήσεις. Ο δεύτερος τριμερής διάλογος θα λάβει χώρα την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου. Αυτά είχα να σας πω όσον αφορά ε, τις ανακοινώσεις. Περνάμε στις ψηφοφορίες. Πρώτη ε, ψηφοφορία. Έχετε έτοιμους τους... Ε, έχετε έτοιμα... Τις κάρτες σας τις έχετε έτοιμες. for agriculture in... Ε, ειδικά μέτρα, πώς, τι είναι, ποια είναι η έκθεση. Ναι, αυτά τα ειδικά μέτρα κλπ. κλπ. Κοινή οργάνωση αγορών αγεωργικών προϊόντων, λοιπόν. Τροπολογία 32, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote Πέρας. Εγκρίνεται. Έχουμε λοιπόν εδώ παρόντες πολιτικές ομάδες, λέει η Πρόεδρος. Αλλάξατε βλέπω τη θέση που καθόσαστε συνήθως και είχα δυσκολία να σας ε, να δω που κάθεστε. Τροπολογία 33 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Block vote από κοινού λοιπόν για τις τροπολογίες 35, 36 και 37 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 38 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 39 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 40 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, ήταν ταυτόσιμη με την τροπολογία 48. Τροπολογία 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Οι 4 και οι 51 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 52 υπέρ κατά η ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 52 άρχεται η, τροπολογία, η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 53 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογίες 54 και 55 από κοινού υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 59 όχι. Φτάνουμε στη συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση. Πολύ ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και εγκρίνεται. Τροπολογία 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 79. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 80. Υπέρ. Α, θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση για την 79. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Τροπολογία 80, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 81, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 82, υπέρ. Κατά αποχέσε, απορρίπτεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 9 και 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 και 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Η ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 110 άρχεται η ψηφοφορία πέρας και εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 112 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 113 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 114 υπέρ. Κατά αποχές ε, ε, το ΕΛΚ ψήφισε, ξαναψηφίζουμε, 114 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 115 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Κυρία Κάντεμπαχ, θέλετε επαλήθευση, πολύ ωραία. Επαλήθευση, ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 115, άρχεται η ψηφοφορία. Ε, ακούστηκε λίγο περίεργα έτσι όπως το είπα για σας, αλλά δεν το εννοούσα. Εγκρίνεται πάντως. 116, τροπολογία 116 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 117 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 118 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 119 υπέρ. Ε, α, ηλεκτρονική επαλήθευση. Κύριε Ντόρφμαν, εσείς ζητήσατε να ελέγξουμε λοιπόν την 118 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. <coughs> Απερίφθη. Τροπολογία 119 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 121 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 124 υπέρ, κατά αποχές το ΕΛΚ ψηφίζει υπέρ ή κατά, υπέρ, άρα εγκρίνεται. Η 124. Τροπολογία 13. Υπέρ κατά αποχές ε, ε απορρίπτεται. 14. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά αποχές Ηλεκτρονική επαλήθευση από τις τροπολογίες 25. Πέρας της ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές. Το ΕΛΚ ψηφίζει υπέρ ή κατά. Ε. Εντάξει, καλύτερα ηλεκτρονική επαλήθευση. γιατί επεκράτησε μια ελαφρά σύγχυση. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 29 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 30 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία πάντα με ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται. Και πέρας και εγκρίνεται. Πολύ ωραία. Περνάμε τώρα στην γνωμοδότηση για το, για το συντονισμό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και συντονισμό της στρατηγικής σχετικά με αυτό. Τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 2 υπέρ αποχές εγκρίνεται, η 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, δεκτή οι σοσιαλδημοκράτες και το ΕΛΚ κατέθεσαν αυτή την τροπολογία. Ας ελέγξουμε λοιπόν, να επαληθεύσουμε την υπαριθμόν 5 τροπολογία. Ήταν ψήφος κατά συνείδηση. Έκλεισε η ψηφοφορία. Ε, δεκτή. Η τροπολογία 6. Υπέρ, κατά, αποχές, το ΕΛΚ είναι υπέρ ή κατά. Δεκτή. Η 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή, η 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή, η 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή, η 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή και τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά ψηφίζουμε παρακαλώ και δεκτό εγκρίνεται το ψήφισμα και έτσι ολοκληρώσαμε ε, τις, ηλεκτρο... τις ψηφοφορίες και τώρα σας καλώ ε, σε μια δημόσια κρόαση ε, για την μείωση των μακροπρόθεσμη και μακροχρόνια μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου αερίων του θερμοκηπίου με βάση και σύμφωνα με την συνθήκη των Παρισίων.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 Αν θέλετε λοιπόν σας παρακαλώ καθίστε ώστε να μπορέσουμε να αρχίσουμε με την ημερησία διάταξή μας δηλαδή με το επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως με μεγάλη μου χαρά σας καλασορίζω όλες και όλους την σημερινή μας ακρόαση για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική και ιδίως τον Επίτροπο και τους έξι ομιλητές που βρίσκονται σήμερα μαζί μας. Όπως γνωρίζετε, στις 28 Ενδεκάτου πέρσι εξέδωσε ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που επιγραφόταν «Καθαρός πλανήτης για όλους». Στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή εξηγεί το μακροπρόθεσμο όραμά τη για μια οικονομία ουδέτερη όσον αφορά το κλίμα μέχρι το 2050. Και εκεί προβλέπει 8 πιθανές πορείες. Η ίδια ανακοίνωση δεν αποτελεί ε, στρατηγική ούτε προσπαθεί να αλλάξει τους συμφωνημένους στόχους του 2030. Προβλέπει επιλογές για δράσεις που θα επιτρέψουν να διεξαχθεί συζήτηση μεταξύ των Ευρωπαίων ε, αξιωματούχων, ηθινόντων κλπ. Για, τον, ε, για την πορεία προς το 2050. Η συζήτηση αυτή θα επιτρέψει στην Ένωση να εγκρίνει και να υποβάλει ε, φιλόδοξη στρατηγική για το 2020 και να καθορίσει την κατεύθυνση για τις μελλοντικέ πολιτικές ενέργειας και κλίματος. Η Επιτροπή μας έχει συμβάλει με δύο προφορικές ερωτήσεις προς Συμβούλιο και Επιτροπή, καθώς και με ψήφισμα. Η ακρόαση εντάσσεται στην συζήτηση που διεξάγει η Επιτροπή μας για το ψήφισμα που παρουσιάζουν, που υποβάλλουν έξι πολιτικές ομάδες και θα συζητήσουμε και μετά το ψήφισμα αυτό, μετά από την ακρόαση. Η ψηφοφορία του ψηφίσματος προβλέπεται για τον επόμενο μήνα με συζήτηση στην Ολομέλεια και ψήφισή τη τον Μάρτιο. Αυτά είναι τα αρχικά μου σχόλια. Κύριε Πίτροπε, σα ευχαριστώ για την προσέλευσή σα Έχετε το λόγο. Ε, αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και εσεί τα μέλη του πάνελ, κυρίε και κύριοι. Σα ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που δίνετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συζητήσει την ανακοίνωσή τη Καθαρό Πλανήτη για Όλου. Ευρωπαϊκή Στρατηγική για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και ουδέτερη για το κλίμα οικονομία, που εγκρίθηκε και υιοθετήθηκε από το Κοινοβούλιο στις 28 Νοεμβρίου 2018. Ευχαρίστως βρίσκομαι πάλι κοντά σα και είμαι ευγνώμων για την ε, ενεργό εμπλοκή του Κοινοβουλίου στη συζήτηση για μια Ευρώπη ουδέτερη ω προ το κλίμα. Με την πρόταση που κάνουμε ανταποκρινόμαστε στην έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να φτιάξει μια στρατηγική μηδενικών εκπομπών για την COP24. Πέρσι και με την ευκαιρία να παρουσιάσουμε μια ε, μακροπρόθεσμη στρατηγική για το πρώτο τρίμηνο του 2018. Ακόμα πιο συγκεκριμένα όμως, η Governance Regulation στο άρθρο 15 υιοθετεί την κυβέρνηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω έχουν κρίνει οι δύο συνομοθέτε, και απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μακροπρόθεσμη στρατηγική, η οποία να εξετάσει τι ενδεχόμενε οδού για να φτάσουμε μέχρι το 2050. Να συμφωνήσουμε τώρα σε μια πορεία για μια ουδετερότητα προς το κλίμα δεν είναι τεχνικό εγχείρημα. Είναι μια ανάγκη στην πράξη. Οι συνέπειε τη αλλαγή του κλίματο είναι ορατέ σε όλη την Ευρώπη. Και πολλοί τα νιώσαμε αυτά και πάνω μα ήδη το καλοκαίρι του 2018. Το μήνυμα των επιστημόνων ε, που ηγούνται των ερευνών ήταν καθαρό στο IPCC, στην δική τους έκθεση για τους 1,5 βαθμούς. Αν δεν δράσουμε τώρα και μάλιστα επιγόντως και συλλογικά τα πράγματα θα χειροτερεύσουν πολύ. Η πολιτική βούληση είναι αναγκαία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το όραμα να δώσει μια ξεκάθαρη πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις προσπάθειές της για το κλίμα και να εντάξει τις ε, συμβολές και την προσπάθεια της αυτή στους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού. Μεγάλη ευθύνη για όλους μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ηγηθούμε παγκοσμίω στην μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και να δώσουμε έτσι και ευκαιρίες για απασχόληση. Έχουμε μια στέρεη αφετηρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των πρώτων στον κόσμο που έχει μια στέρεα νομοθεσία για το 2030, η οποία θα επιτρέψει να υλοποιήσουμε τις υποσχέσεις μας αυτό, για να συμφωνήσουμε πάνω σε αυτό δεν ήταν εύκολο. Χάρη στη σκληρή δουλειά, αποφασιστικότητα και επικοδομητικότητα, και αναγνωρίζω εδώ βεβαίω και το σημαντικό ρόλο τη της ε, Επιτροπή σα και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα καταφέραμε. Ακόμα καλύτερα. Η πλήρη εφαρμογή στην επόμενη δεκαετία τη νομοθεσία για το κλίμα και την καθαρή ενέργεια θα μα επιτρέψει να μειώσουμε τι εκπομπέ μα κατά 45% μέχρι το 2030 σε σύγκριση με το 1990, το οποίο θα σημάνει ότι έχουμε επιτύχει de facto τον στόχο μας του 2030 για 40%. Για να συμβεί όμως αυτό, η νομοθεσία πρέπει πρωτίστως να ακολουθείται από ρωμαλαίες δράσεις επιτόπου. Οι χώρες μέλη έχουν κάνει το πρώτο βήμα και η πλειοψηφία τους έχουν υιοθετήσει εθνικές πολιτικές και μέτρα στα σχέδια των εθνικών, ε, μάλλον στα εθνικά σχέδια για το κλίμα και την ενέργεια. Αλλά για να είμαστε σαφείς, οι πολιτικές με το 2030 θα καλύψουν μεγάλο έδαφος. Οι στόχοι του 2030 ήδη βρίσκονται στο στάδιο της μετάβασης και θα απαιτήσουν σημαντικές αυξήσεις σε μακροπρόθεσμες παραγωγικές επενδύσεις. Χρειάζεται όμως ακόμα περισσότερη δράση. Οι προσπάθειές μας μέχρι το 2030 θα πρέπει να υπερβούν και το 2030 θα οδηγήσουν όμως μόνο σε 60% μειώσεις των εκπομπών το 2050, το οποίο δεν αρκεί για να συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού. Γι' αυτό και θα πρέπει να ενισχύσουμε τις πολιτικές πέραν του 2030 και οποιασδήποτε εξελίξει πολιτικής στο μέλλον θα πρέπει να λάβουν την εικόνα μετά το 2030 υπόψη τους. Να έρθω τώρα στο, στο μακροπρόθεσμο όραμα και να σας δώσω τις βασικές γραμμές του. Πρώτον, σε ό,τι αφορά το επίπεδο φιλοδοξίας. Προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθεί προς μια ουδετερότητα σε ό,τι αφορά το κλίμα, δηλαδή μηδενικές εκπομπές ρίων θερμοκηπίου μέχρι το 2050. Αυτό είναι το επίπεδο φιλοδοξίας το οποίο θα πρέπει να επιδιώξει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιτύχει τους στόχους του 1,5 βαθμού των Παρισίων. Από την άλλη μεριά, η σε βάθος ανάλυσης δείχνει ότι για να διατηρηθεί βιώσιμη ανάπτυξη, δουλειές και βελτιωμένη ποιότητα τη ζωή των πολιτών απαιτούνται αυτέ οι κινήσει. Αυτή η ανάλυση βασίζεται σε μοντέλα τα οποία προέρχονται από διάφορου ενδιαφερομένου και ερευνητικέ μελέτε, μεταξύ αυτών και την έκθεση τη IPCC για τον 1,5 βαθμό. Πέρα αυτού, θεωρούμε τα απορίσματα τη δημόσια διαβούλευση τα οποία έχουμε λάβει από μεγάλο, βαθμό, από μεγάλο αριθμό μάλλον ενδιαφερομένων που μας επιτρέπει να διακρίνουμε 8 σενάρια με διαφορετικά επίπεδα φιλοδοξίας αλλά όλα εντός των πλαισίων της Συμφωνίας του Παρισιού. Πέντε από τα σενάρια αυτά στοχεύουν σε μείωση κατά 80%, μία κατά 90% και δύο αξιολογούν την επιλογή μηδενικών εκπομπών που είναι συμβατή με τον στόχο της, του περιορισμού της αναθέρμανσης του κλίματος σε 1,5 βαθμό έως το 2050. Πρέπει να αναλύσουμε όλες αυτές τις τεχνολογίες και τις ενδεχόμενες λύσεις, ηλεκτροκίνηση, υδρογόνο, ε, συνθετικά αέρια και κυκλική οικονομία. Εάν συνδυαστούν αυτά και με ισχυρή συμβολή από, την, ε, από τους άλλους τομείς, τα αποτελέσματα θα είναι ικανοποιητικά μέχρι το 2050. Δεύτερο, για το πώς θα φτάσουμε εκεί χρειάζονται ορισμένες επιλογές που να είναι στέρεες και να επιτρέψουν την υιοθέτηση αυτών των σενάριων. Σε όλες τις ε, ε, επιλογές που αναλύουμε, τα συστήματα ενέργειας βασίζονται σε μια ασφαλή και βιώσιμη παροχή ενέργειας. Με αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και με χρήση ε, ανανεώσιμων πηγών. Στο μέλλον θα χρειαστούν αυτά για να μπορέσουμε να μειώσουμε την κατάλληλη ενέργειας στο μισό σε σύγκριση με το 2005. Σήμερα το 40% της κατανάλωσης ενέργειας είναι από τα κτίρια. Τα περισσότερα από τα κτίρια υπάρχουν ήδη, άρα θα πρέπει να τα ανακαινιστούν. Στα μέσα του αιώνος θα υπάρξει παντού ηλεκτροδότηση και το ηλεκτρικό ρεύμα θα διπλασιάσει την χρήση του. Πάνω από 80% του ηλεκτρικού ρεύματο θα προέρχεται από ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και θα χρειαστούν και άλλα σχετικά μέτρα. Η ουδετερότητα σε ό,τι αφορά το κλίμα δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρί ένα σύστημα καθαρή κινητικότητα. Η ηλεκτροκίνηση είναι σαφώ ο δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Αλλά θα χρειαστούν και άλλα μοντέλα ε, μεταφορών. Το να μπορέσουμε τώρα ε, να χρησιμοποιήσουμε και το δυναμικό της βιοοικονομίας είναι επίσης ένα σημαντικό, ένα κεντρικό, ένας κεντρικός στόχος. Εδώ θα χρειαστούμε όμως να βρούμε μια ισορροπία. Γεωργία και δασοκομεία μπορούν να βοηθήσουν στο να απαλλαγούν από τα διοξίδια του άνθρακα ή άλλοι τομείς της οικονομίας. Αλλά πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας ώστε θα κάνουμε την καλύτερη δυνατή χρήση του, του, των διαφόρων φυσικών πόρων για να μειώσουμε και τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακο που δεν μπορούμε να μειώσουμε διαφορετικά. Με την ανάπτυξη τη ανανεώσιμη ενέργεια, αυτή δεν είναι πανάκια, παρόλα αυτά παίζει σημαντικό κρίσιμο ρόλο για την αντιμετώπιση των υπόλοιπων εκπομπών από βιομηχανίε ε, εντατικέ στη χρήση ενέργεια. Για να γίνουν αυτά τα πράγματα χρειάζεται και κοινωνική εμπλοκή και μια δίκαιη μετάβαση, στοχευμένη χρηματοδότηση, έρευνα και ανάπτυξη, αλλαγές στη συμπεριφορά των πολιτών. Για να γίνει η μετατροπή αυτή χρειάζεται να λάβουμε υπόψη, για παράδειγμα, ότι χρειάζεται να λάβουμε υπόψη και τις επιπτώσεις στην οικονομία και στην απασχόληση. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και συλλογική δράση. Κανένας δεν μπορεί να μείνει πίσω. Θα πρέπει λοιπόν να είναι οι προσπάθειες αυτές να μην αποκλείουν κανένα και να είναι κοινωνικά δίκαιες η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρε μέλη να αναπτύξουν όλε τι σωστέ πολιτικέ για να αντιμετωπίσουν την πρόκληση. Δημοσιονομική πολιτική, πολιτική απασχόληση, πολιτική συνοχή, όλε έχουν να παίξουν ένα ρόλο για να μειωθούν οι ε, αποκλήσει οικονομικέ και ταφικέ σε ολόκληρη την Ένωση. τα, τα διάφορα ε, ε, πιλωτικά προγράμματα επίση πρέπει να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο. Προτιθέμεθα να ξεκινήσουμε μια συμπεριληπτική και ενημερωμένη συζήτηση μεταξύ Ευρωπαίων πολιτών, ενδιαφερομένων μερών και όσων λαμβάνουν τις πολιτικές αποφάσεις. Τα επόμενα βήματα, φέτος το 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διεξαγάγει σημαντικές δραστηριότητες για να προσεγγίσει τους ενδιαφερομένους και εντός και εκτός Ευρώπης. Αναμένω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει ψήφισμα για το μακροπρόθεσμο όραμα στους επόμενου μήνες και αναμένω την ενεργό εμπλοκή του και τον υπόλοιπο χρόνο η ομάδα μου και εγώ θα αρχίσουμε να επισκεπτόμαστε τις χώρες μέλη ήδη από τον επόμενο μήνα. Θα χρειαστούμε ευρύτατη υποστήριξη από όλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αρχίσει να συζητεί τα θέματα αυτά στα διάφορα συμβούλια και η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, θα προσφέρουν τις αναγκαίες κατευθυντήριες γραμμές. Αναμένω λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον την καρποφόρο συζήτηση σήμερα, αλλά και βεβαίως σε όλο το 2019. Σε ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ και επίτροπε για την ε, παρουσίασή σας. Και τώρα θα παρακολουθήσουμε τις ε, παρουσιάσεις των ε, προσκεκλημένων μας του πρώτου πάνελ. Θα ακολουθήσει συζήτηση και μετά θα περάσουμε στο δεύτερο πάνελ. Για το πρώτο χαίρομαι που έχω, το, έχω την δυνατότητα να καλωσορίσω τον πρόεδρο της COP24 και ο οποίος είναι και υφυπουργός τη Δημοκρατία τη Πολωνία, υπουργό περιβάλλοντο, ο κύριος Μίχαλ Κούρτικα. Έχετε το λόγο κύριε. Thank you very much, ladies and gentlemen. Ευχαριστούμε πολύ κυρίες και κύριοι. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά για μένα που μπορώ να βρίσκομαι εδώ στις Βρυξέλλες. Ε, κύριε Πίτροπε, χαίρομαι πολύ ε, που μπορώ να λάβω το λόγο μετά από εσάς. Με αυτή τη ε, συζήτηση θα ήθελα να σας πω λιγάκι τι κάναμε στην Κατοβίτσα από κοινού με τον Επίτροπο. Δηλαδή συζητήσαμε για τη Συμφωνία του Παρισιού και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για την επιτυχία και βεβαίως ε, είναι ε, σημαντικά ε, τα θεμέλια που τίνεται εδώ στην Ευρώπη για το μέλλον της περιβαλλοντικής πολιτικής. Πρώτα απ' όλα θα πω λίγα λόγια σχετικά με την συμφωνία COP24, τη διάσκεψη των συμβαλωμένων μερών, την 24η. Είναι δύσκολο να επιτύχει κανείς σε μια συμφωνία ανάμεσα σε όλα τα μέρη ε, τη Συμφωνίας του Παρισιού, αλλά τα καταφέραμε. Ε, μπορέσαμε όλοι από κοινού να βρούμε έναν τρόπο έτσι ώστε να περάσει αυτή η συμφωνία και να μπορέσουμε ε, να δώσουμε ζωή και πάλι στην ε, διεθνή αλληλεγγύη. Και λέω και πάλι γιατί ζούμε σε μια ιδιαίτερα ε, πολυτάραχη πολιτική και γεωπολιτική κατάσταση και αυτό που μπορούσε να γίνει το 2015 στο Παρίσι ήταν πολύ πιο δύσκολο μετά από τρία χρόνια στην Κατοβίτσα. Χωρίς λοιπόν την βούληση όλων να, κάνουν, να επιτύχουν μια συμφωνία και να ε, βρεθούν σε αλληλεγγύη με τους άλλους, ήταν δύσκολο να καταλήξουμε σε συμβαστική λύση. Και βεβαίως αυτό προσφέρει και την ε, ασφάλεια, την νομική για την παγκόσμια πολιτική για το κλίμα, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο μετά ε, το ότι το 2020 θα εκπνεύσουν οι κανόνες που συμφωνήθηκαν στο Κιώτο. Από το 2021 θα αρχίσει να ισχύει η Συμφωνία του Παρισιού και ε, μετά την Κατοβίτσα μπαίνουμε πλέον σε μια διαφορετική εποχή των παγκόσμιων κανόνων για το κλίμα. Τώρα κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν γνωρίζει πώς να εφαρμόσει τη Συμφωνία του Παρισιού. Και κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί τι ακριβώς σημαίνει να ε, προσφέρει ε, τις ε, δυνατότητες για να ολοκληρωθούν οικουμενικές προσπάθειες. Εμείς στην Κατοβίτσα συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα κεφάλαιο το οποίο να έχει σχέση με τη μείωση των εκπομπών. Εξάλλου μπορεί να υπάρχουν και άλλα στοιχεία όπως είναι η προσαρμογή ή κάποιες διατάξεις για τη χρηματοδότηση. Έχουμε λοιπόν τους κανόνες της Κατοβίτσα. Έχουμε επίσης το πλαίσιο ε, Και νομίζω ότι αναμφίβολα το βασικότερο επίτευγμα της COP24 είναι αυτό που ε, ακριβώς ανέφερα, δηλαδή συμβιβασμός και λεπτομερείς ε, κανόνες για τη Συμφωνία του Παρισιού. Αυτός είναι ο ε, κοινός παρανομαστής που αφορά όλα τα μέρη. Εργαστήκαμε λοιπόν με όλους τους υπουργού που έρχονται από αναπτυγμένες αλλά και αναπτυσσόμενες χώρες. Μπορέσαμε να επιτύχουμε ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα με κοινούς κανόνες για όλες τις χώρες αλλά και με οικονομική βοήθεια και ευελιξία για εκείνες τις χώρες που χρειάζονται τη βοήθεια. Να είμαι όμως απόλυτα σαφές. Ε, συγκλίνουμε προς ε, ένα σύστημα διαφάνειας και αυτό είναι κάτι που το θεωρώ πολύ σημαντικό. Το πετύχαμε στην Κατοβίτσα. Δουλεύουμε ε, με τους συναδέλφους μας από την COP25 για να ολοκληρώσουμε άρθρο όπως είναι αυτό το άρθρο 6 ε, που έχει σχέση με την αγορά ε, διοξιδίου του άνθρακα. Η Πολωνική Προεδρία πρότεινε επίσης ε, να δουλέψει για την ε, τεχνολογία και την ανθρώπινη φύση και κάθε ένα από αυτά εκφράστηκε με τη μορφή δήλωσης. Αρχίσαμε λοιπόν την πρώτη μέρα της COP ε, με την ε, αλληλεγγύη, την δήλωση για την αλληλεγγύη και την δικαιοσύνη. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ήταν στην αρχή της συνδιάσκεψης ε, που ξεκίνησε με την Πολωνική Προεδρία, όπου παρίστατο και ο κύριος Αντιόνα ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Όσον αφορά αυτή τη δίκαιη μετάβαση, αυτό ήταν ένα συμβολικό ε, εργαλείο με την έννοια ότι η COP24 έλαβε χώρα στην Κατοβίτσα ε, που είναι ε, πρωτεύουσα μιας περιοχής με περίπου 5 εκατομμύρια ανθρώπους. Ε, είναι μια περιοχή βαριάς βιομηχανίας, εξορίξεων. Τώρα εκεί γίνονται πολλές αλλαγές. Έχουμε μικρή ανεργία, έχουμε μεγάλη συγκέντρωση νέων υπηρεσιών, άρα δηλαδή είναι επιτυχημένο παράδειγμα αλλαγής. Είπαμε επίσης ότι είναι απαραίτητο να ε, υπάρχει ε, εξισορρόπηση ε, για τις εκπομπές ε, που εκλείονται. Γνωρίζουμε ότι αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για τη βιοπικιλότητα και για την ποιότητα ζωής μας. Και τέλος, αποδώσαμε σημασία στο γεγονός ότι αρχίζουμε να έχουμε τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν ως προς την επίτευξη των ε, κλιματικών μας ε, στόχων. Βέβαια θέλουμε να έχουμε και βιομηχανικά ωφέλη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια χώρα όπως είναι η Πολωνία. Γιατί εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα που έχουν σχέση με την ατμοσφαιρική ρήπανση. Γι' αυτό λοιπόν ο εξηλεκτρισμός ε, των μεταφορών είναι βασικός στόχος για την Πολωνία. Και για να επιτευχθεί αυτό ε, δημιουργούμε ένα στόλο ηλεκτρικών λεωφορείων και έχουμε και έναν φιλόδοξο στόχο για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτά ε, είναι πολύ σημαντικά για χώρες ε, όπως η Κίνα, η Ινδονησία, ε, αλλά και η Ιαπωνία, η Κορέα, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία. Κατά κάποιον τρόπο όλα αυτά είναι και συμβολικά, γιατί αρχίζουμε να έχουμε συγκεκριμένες τεχνολογίες οι οποίες ε, αρχίζουν ε, να ε, οδηγούν στην υλοποίηση του οράματος το οποίο παρουσίασε ο Επίτροπος κ. Κανέτε. Ένα μήνα μετά την Κατοβίτσα. Εδώ βρισκόμαστε τώρα. Έχουμε ένα νομικό πλαίσιο για την ε, ε, για την περιβαλλοντική πολιτική, έχουμε και τη Συμφωνία όλων των κρατών μελών και έχουμε ε, και ένα νομικό πλαίσιο μέχρι το 2030. Αυτό που πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι να υπάρχει η εφαρμογή και η εστίαση στην εφαρμογή, στην επίτευξη των στόχων, αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Άρα δηλαδή χρειαζόμαστε όχι μόνο τεχνολογίες, νομίζω για πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε την απαραίτητη τεχνολογία, αλλά εκείνο που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό είναι και ότι χρειαζόμαστε κοινωνική αποδοχή, ε, χρειαζόμαστε κοντά μας ε, τις κοινωνίες, όχι ενάντια σε μας, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας, τις φιλοδοξίες μας. Ε, πρόκειται λοιπόν να εφαρμόσουμε όλες αυτές τις ε, στρατηγικές. Ελπίζω να έχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα ε, και μετά ο πρώτος απολογισμός θα γίνει με βάση τους νέους κανόνες το 2023. Τώρα, αναφέρομαι στο τελευταίο στοιχείο, το οποίο έχει σχέση με τη μακροχρόνια στρατηγική ξεκινήσαμε αυτή τη συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλα αυτά δεν συνδέονται πλέον μόνο με την ενέργεια, αλλά και με άλλους τομείς, με τις ε, μεταφορές. Ε, εκεί υπάρχουν πάρα πολλές ε, δυσκολίες. Έχουμε την μεγαλύτερη αύξηση εκπομπών σε χώρες του ΟΣΑ. Εκεί είναι η μεγαλύτερη αύξηση στον τομέα των μεταφορών. Γι' αυτό πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να μετατρέψουμε τον τομέα αυτό. Αυτό που παίζει ρόλο είναι επίσης και τα κτίρια. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν εδώ ε, θα έχουν πρακτικές συνέπειες όχι μόνο για μετά από 10-20 χρόνια, αλλά και μετά από 50 χρόνια. Ε, είναι λοιπόν πολύ περίπλοκο το να αντιμετωπιστεί και το θέμα των εκπομπών στη Γεωργία. Ως εκ τούτου, η ε, Πολωνία δουλεύει σκληρά σε όλα αυτά. Ε, θέλουμε να εξισορροπήσουμε ε, τις εκπομπές ε, όπως αναφέρθηκε και η Συμφωνία του Παρισιού η μακροχρόνια στρατηγική είναι ευπρόσδεκτη ε, και τώρα έχουμε αρχίσει να σκεφτόμαστε κατά πόσον είναι γενικότερα δυνατό να έχουμε κάποια συγκέντρωση ενέργειας να συγκεντρώσουμε και προγράμματα για την κλιματική αλλαγή από τα κράτη-μέλη, ε, να καταλήξουμε δηλαδή σε κάτι ε, το οποίο θα ικανοποιεί όλους μας. Νομίζω ότι αυτή η φιλοδοξία απαιτεί ε, πολλές επενδύσεις και αυτή τη στιγμή κοιτάμε λίγο τον μέσο όρο, κοιτάμε μεσοσταθμικά τις επενδύσεις, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε ε, ποιες χώρες μπορούν να στηρίξουν, να αναλάβουν αυτό το βάρος. Ε, πόσο γρήγορα μπορούν να προχωρήσουν οι διάφορες χώρες και νομίζω ότι ε, η ταχύτητα θα ποικίλει. Δηλαδή θα υπάρχουν χώρες οι οποίες θα είναι σε θέση να φτάσουν στο σημείο εκείνο που ανέφερε και ο κύριος Κανιέτε την ουδετερότητα ως προς το κλίμα. Κάποιες χώρες θα την επιτύχουν νωρίτερα, αλλά άλλες έχουν μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα, θα χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Ε, χρειαζόμαστε, ε, πρέπει να σκεφτόμαστε με αλληλέγγυο τρόπο για να επιτύχουμε την ουδετερότητα ως προς το κλίμα η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα πρέπει να λάβει υπόψη τις διάφορες καταστάσεις που επικρατούν ε, στα κράτη-μέλη, διαφορετικά σημεία κίνησης. Νομίζω ότι το 2020 ε, το 19 μάλλον θα είναι σημαντικό για μας, για να σκεφτούμε το μέλλον μας, αλλά και για να σκεφτούμε για την Προεδρία COP24, που θα συμμετέχει εργα, ενεργά στη συνάντηση κορυφής ε, του, των Ηνωμένων Εθνών που θα λάβει η χώρα το Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη. Και εκεί θα τεθεί και το θέμα ε, του πώς συζητάμε για τους ε, οικουμενικούς παγκόσμιους στόχους. Και παράλληλα βέβαια θα πρέπει να προχωράει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, ο επόμενος ομιλητής είναι ο, Γενική, ο Γενικός Διευθυντής της της Ευρωπαϊκής Σημικής Βιομηχανίας. και εκπροσωπεί 11 κύριους τομείς. Είναι μέρος της ΕΣΠΑ. Thank you, Madam Chairman. Thank Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ που μας δώσατε τη δυνατότητα να μιλήσουμε σήμερα εξ ονόματος της βιομηχανίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκπροσωπώ την ΣΕΦΙΚ, αλλά σήμερα εδώ ε, εκπροσωπώ την ΣΠΑΡΙΑΡ που είναι ε, η σύμπραξη ιδιωτικού δημοσίου τομέα ε, για τα χημικά, για το ρέμιξ για το, και για άλλους βιομηχανικούς τομείς τομείς. Ε, χαίρομαι που μπορώ να μιλήσω εδώ, ε, γιατί ε, εμείς προσπαθήσαμε μέσω μιας έκθεσης που αφορούσε ακριβώς την απελευθέρωση της Ευρώπης από τον άνθρακα. Συμβάλαμε, λέω, μέσω αυτού στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, πολλά από τα στοιχεία της δουλειάς μας αναφέρονται και στο Staff Working Document της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Ε, θέλαμε γι' αυτό να ευχαριστήσουμε ε, και τον Επίτροπο και την υπηρεσία του, καθώς επίσης και τη Γενική Διεύθυνση GROW. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι ε, να ε, δείξουμε τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε και τι ακριβώς μπορεί να περιμένει κανείς από εμά και θα ήθελα να πω δύο λόγια σχετικά με αυτά. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα μείγμα καινοτόμων ε, τεχνολογιών. Ε, όσον αφορά την δέσμευση και αποθήκευση και χρήση του άνθρακα, ε, το CCS ε, για τις εκπομπές τις οποίες δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε διαφορετικά. Η κυκλική οικονομία θα συγχωνευτεί με την χαμηλών εκπομπών άνθρακα οικονομία και οι μελέτες δείχνουν κυρίως ας πούμε για την χημική βιομηχανία ότι η ανακύκλωση των χημικών υπολείπων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλά έγιναν τα προηγούμενα δέκα χρόνια, αλλά τα επόμενα δέκα χρόνια είναι πολύ αποφασιστικής σημασίας ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε κάποια εμπορικά στοιχεία τα οποία να είναι πολύ ε, ε, σημαντικά. Εμείς ε, δουλεύουμε σαν βιομηχανία έτσι ώστε να προχωρήσουμε και να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αλλαγές. Η ανάγκη για ηλεκτρισμό και η χρήση επομένως των ανανεώσιμων πηγών είναι πολύ μεγάλης σημασίας. Βεβαίως οι υπολογισμοί γίνονται λίγο με διαφορετικό τρόπο από την Κομισιόν και από εμά. Ωστόσο, στον χάλιβα ε, για τον άνθρακα και για τον ε, χάλιβα ε, θα χρειαστούμε τέσσερις με πέντε φορές τις ανάγκες σε ηλεκτρισμό της γερμανικής ε, βιομηχανίας. Επομένως καταλαβαίνετε ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικές οι προσπάθειες που πρέπει να γίνουν και πολύ μεγάλες οι απαιτήσει σε ηλεκτρισμό. Θα πρέπει να καθορίσουμε το στόχο, να ταυτοποιήσουμε τις ε, τεχνολογίες, να δούμε τα πιλωτικά προγράμματα, αλλά βεβαίως η δυσκολία έγκυται ε, στην εξέβρεση των πραγματικών προγραμμάτων και τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι νέες ε, τεχνολογίες. Ε, εδώ χρειάζεται αυτή η παγκόσμια ε, διαδικασία. Θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε τι θα κάνουμε με τις εισαγωγές και οπωσδήποτε οι εισαγωγές-εξαγωγές να βρίσκονται ακριβώς στο ίδιο επίπεδο και να έχουν την ίδια μεταχείριση αν θέλουμε να σώσουμε τις αγορές. Εμείς θεωρούμε ότι η ενσωμάτωση των τομέων αποτελεί την προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία και θεωρούμε ότι και στον, ε, στον τομέα των χημικών, ας πούμε, το υδρογόνο μπορεί να αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα. Χρειαζόμαστε όμως υποδομές. Ε, αυτή τη στιγμή ε, είτε είναι πολύ περιορισμένη η εικόνα, ε, είτε πρέπει να αποσαφινιστεί περαιτέρω η εικόνα. Χρειαζόμαστε διασυνδέσεις μεταξύ των αγωγών και ανάμεσα στο αίτιασα και το Ταμείο της Καινοτομίας, ανάμεσα ε, στα, στις επενδύσεις και τα διαφορετικά ταμεία θα πρέπει να βρεθεί ο κοινός τόπος που θα οδηγήσει σε αύξηση των επενδύσεων. Αυτό που χρειάζεται είναι και αυτό που εμείς ονομάζουμε master plan ε, για την ε, ε, τροποποίηση, για την αλλαγή της βιομηχανίας. Χρειαζόμαστε πραγματικά ένα τέτοιο master plan, το οποίο θα μετακινήσει την ανάγκη να αναλάβει και η βιομηχανία πρέον το ρόλο που πρέπει. Συζητούμε τα θέματα αυτά με εκπροσώπους της Κομισιόν και κάποιος αστιαβόμενος είπε «Ποτέ δεν θα έχετε βιομηχανική πραγματική πολιτική μέχρι ότου ε, ο ε, μέχρι ότου να υπάρχει ένας ε, αντιπρόεδρος της ε, Κομισιόν που θα αποδίδει στον Επίτροπο Περιβάλλοντος και στον Επίτροπο Ανταγωνισμού και στον Επίτροπο Εμπορίου. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει μία σύνδεση όλων αυτών πρέπει οπωσδήποτε να δούμε και ποιος είναι ο, ο χώρος που καταλαμβάνει και πρέπει να καταλαμβάνει η βιομηχανία, καθώς επίσης ε, ε, και αυτή η ε, απόρρια τεχνολογίας μέσω ντέμος και πιλωτικών, αλλά πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οπωσδήποτε στην ευρεία εμπορική διάσταση γίνονται επενδύσεις. Εσείς ζητάτε κάποια ζητήματα στην γνωμοδότησή σας. Πρώτα απ' όλα αναφέρεστε σε βιομηχανία χαμηλών εκπομπών άνθρακα ε, και ε, τα ε, οπωσδήποτε θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα JTI για το υδρογόνο, τα IPCIs, ε, οι συμπράξεις αυτές ε, του Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και οπωσδήποτε θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και από την επόμενη Επιτροπή και από την παραπέρα Επιτροπή. να υπάρχουν δεσμευτικοί στόχοι για την Ευρώπη και λέμε ότι θα πρέπει εμείς να ε, είμαστε σαν βιομηχανία αυτό το καναρίνι το οποίο καταφέρνει και ζει παρά τις, ε, τα αέρια που εκλείονται στο ορυχείο οπωσδήποτε αναδιάρθρωση και ανασχηματισμό της, ε, ε, της νομοθεσίας έτσι ώστε η κυκλική οικονομία να διασυνδεθεί με την χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Ε, επίσης ε, διασύνδεση των διαφόρων τομέων της βιομηχανίας, πράγμα που προαπαιτεί βεβαίως αλλαγή, αλλαγές, ε, πράγμα που προϋποθέτει επίσης και αλλαγή των υποδομών καθώς επίσης και της προμήθειας άνθρακα που χρειάζεται ε, η βιομηχανία για να επιβιώσει. Εμείς ε, συνεργαζόμαστε και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την Κομισιόν γιατί θέλουμε να παίξουμε το ρόλο που μας αρμόζει σε αυτήν την μετάβαση αλλά θέλουμε η μετάβαση να γίνει σωστά στην ε, Ευρώπη. Θέλουμε τα υλικά να γίνονται στην Ευρώπη, να διατίθενται στην Ευρώπη ε, η μεταποίησή τους να λαμβάνει χώρα στην Ευρώπη. Εν συμπεράσματι νομίζω ότι είναι επικοδομητική η θέση της βιομηχανίας, τα στοιχεία υπάρχουν αλλά χρειαζόμαστε και έναν επικοδομητικό τρόπο συνεργασίας για να προχωρήσουμε στην επόμενη δεκαετία, έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι οι επενδύσεις θα γίνονται και θα μένουν στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μένσινγκ. Ο κύριος Μπεζαμέν Ντενή, ο οποίος είναι σύμβουλος για την ενέργεια και το κλίμα ε, στην ε, ΕΤΟΚ, ε, στην Συνομοσπονδία, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους σας. Ε, η Συνομοσπονδία Συνδικάτων είναι μια συνομοσπονδία η οποία εκπροσωπεί 90 ε, συνδικάτα τα οποία έρχονται από, τις, ε, από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ε, εμείς πραγματικά καλωσορίζουμε την μακροχρόνια στρατηγική, το σχέδιο εγγράφου το οποίο δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα γιατί πιστεύουμε ότι το έγγραφο αυτό ταιριάζει καλύτερα με τις ε, φιλοδοξίες μας ε, ε, και με την επιστήμη. Μετά από πολλές και δημοκρατικές συζητήσεις με τα μέλη μας, επίσημα υιοθετήσαμε ως βασικό στόχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση την ανάγκη να υπάρχουν μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, σε μια οργάνωση η οποία εκπροσωπεί τους εργαζόμενους από όλους τους τομείς και από όλα τα κρατη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό είναι πρόκληση. Παρά όμως ε, τις ε, διαφορετικές απόψεις που μπορεί να υπάρχουν για τη σηματοδοχή υπάρχει ε, και κάποια ισχύει το κατεπήγον και πρέπει οπωσδήποτε να δράσουμε. Έτσι λοιπόν φτάνω στην πρώτη μου επιφύλαξη ε, σχετικά με τη μακροχρόνια στρατηγική όπως αυτή δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή. Εάν ο στόχος της μακροχρόνιας στρατηγικής είναι να ε, εμπνεύσει και να κατευθύνει τις δράσεις, δεν καταλαβαίνουμε γιατί ευθύς εξ αρχής κρίνεται ότι όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα των διαφόρων υπολογισμών, δεν θα μπορέσουμε να επανεξετάσουμε ε, τους στόχους του 2020. Δηλαδή, αν ήδη γνωρίζουμε ότι τα νυν εργαλεία της πολιτικής δεν θα μπορέσουν να προσφέρουν αυτά που ζητάει η επιστήμη και που είναι και οι στόχοι του Παρισιού, τότε γιατί τα διατηρούμε όλα αυτά. Εμείς ως συνδικάτα δεν θέλουμε ε, να μπούμε και σε άλλον ένα, σε μια δεκαετία με μηδέν μέτρα. Ε, θεωρούμε ότι πρέπει κάτι να γίνει, να αναλάβουμε δράση ε, και θεωρούμε ότι οι άνθρωποι που περπατούν ε, στους δρόμους ε, ακριβώς αυτό θέλουν. Εξάλλου χαιρετίζουμε τη μακροχρόνια στρατηγική γιατί προσφέρει και πολύ καλύτερη ανάλυση της κοινωνικής διάστησης της διαδικασίας απομάκρυνσης του άνθρακα δείχνουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν ε, σε τομείς όπως είναι οι κατασκευές, οι, οι ε, πράσινες θέσεις απασχόλησης, ανανεώσιμη ενέργεια και εντοπίζεται μία σειρά ε, πολύ σοβαρών και συγκεκριμένων προκλήσεων όσον αφορά την ε, απασχόληση σε τομείς ε, όπου τα ωφέλη της οικονομίας ε, χαμηλής χρήσης άνθρακα είναι πολύ πιο δύσκολο να διασφαλιστούν. Εξάλλου, καθίσατε σαφές πως όλες αυτές οι προκλήσεις αφορούν όλες τις περιοχές και τα κράτη-μέλη. Ειλικρινά, καλωσορίζουμε αυτό το γεγονός και θεωρούμε ότι αποτελεί πολύ μεγάλη πρόοδο σε σχέση με το χάρτη πορείας ε, μέχρι το 2050. Ε, χαιρετίζουμε επίσης το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες ε, πρωτοβουλίες όπως η πλατφόρμα COP σε μετάβαση, αυτές οι πρωτοβουλίες θα στεφτούν από επιτυχία. Υπάρχει το εξής. Αυτή η στρατηγική παρουσιάζει ένα είδος ε, ολοκληρωμένης ε, βιομηχανικής πολιτικής ε, περιορισμένης χρήση του άνθρακα. Θα σας εξηγήσω γιατί απομένουν κάποιες, κάποια ερωτήματα, αλλά είμαστε πολύ πιο μακριά πλέον από την αμυντική στάση που είχαμε εδώ και πολλά χρόνια. Με βάση δηλαδή βραχυπρόθεσμους ορισμούς της ανταγωνιστικότητας. Τώρα έχουμε ένα πολύ καλό μείγμα ε, καινοτόμων ε, ε, επιθετικών εργαλείων. Όπως σας είπα λοιπόν, εξακολουθούν να υπάρχουν ανοιχτά κάποια ερωτήματα που θέλουμε να θίξουμε. Έχουμε κάποιες ανησυχίες το πρώτο θέμα που θέλω να δείξω έχει σχέση ε, με τις ε, τεχνολογίες χαμηλής χρήσης του άνθρακα. Στο χάρτη πολύ αναφέρεται ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει μέχρι το 2050 να είναι ουδέτερη ως προς τη χρήση άνθρακα, πρέπει ταχύτατα να αναπτύξει μία σειρά τεχνολογιών χαμηλής χρήσης άνθρακα για να απομακρυνθεί ο άνθρακας από αρκετούς τομείς και εκεί πρέπει να υπάρξουν καινοτομίες. Αυτό δεν είναι κάτι το καινούριο. Γνωρίζουμε εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια ότι είναι απαραίτητο να υπάρξουν νέες τεχνολογίες. Αν πάρουμε τη δέσμευση και τη αποθήκευση του άνθρακα, το CCS, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή την τεχνολογία την έχει χαρακτηρίσει ως βασική ε, για να απομακρυνθεί ο άνθρακας. Ε, δέκα χρόνια αργότερα δεν υπάρχει όμως ε, καμία βιομηχανία κλίμακας ε, με αυτήν την τεχνολογία που να λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ρωτώ γιατί. Γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση ως προς το να εφαρμόζονται αυτές οι τεχνολογίες. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε στο έγγραφο της Κομισιόν είναι ότι θα συνεχίσει η Κομισιόν να κάνει αυτά που κάνει εδώ και τα τελευταία δέκα χρόνια. Δηλαδή ε, να ε, διασφαλίζει προϋπολογισμούς ε, και κονδύλια για την καινοτομία. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι υπάρχει μία απόσταση ανάμεσα στην αίσθηση του κατεπήγοντος που αναφέρεται στο έγγραφο και εντάξει, μερικοί λένε έχουμε άλλε τρει δεκαετίε για να απομακρυνθεί πλήρως ο άνθρακας από την οικονομία. Από την άλλη υπάρχουν κεφάλαια που αφορούν τη βιομηχανική καινοτομία και εκεί αναφέρεται ότι θα προσπαθήσουμε να ε, κινητροδοτήσουμε την ε, τεχνολογία μέσα από κάποια χρηματοδοτικά προγράμματα. Ε, εμείς ε, δεν πιστεύουμε ότι αυτή η ασάφεια συμβαδίζει με την αίσθηση του κατεπήγοντος. Ε, και πάλι χρειαζόμαστε ενημερωτικές πολιτικές μεταρρυθμίσεων που θα διασφαλίζουν νέες τεχνολογίες για την απομάκρυνση του άνθρακα. Αυτές οι τεχνολογίες να εφαρμοστούν έγκαιρα και όπως βλέπετε ο στόχος μας δεν είναι να πούμε εμείς ποια είναι η καλύτερη τεχνολογία για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Εμείς απλά θέλουμε να αναφέρουμε ότι αυτές οι τεχνολογίες δεν έχουν ακόμα ε, χρησιμοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ ίσως μπορούμε να ανοίξουμε θέματα τα οποία δεν ανοίγουν ακόμα στο έγγραφο. Όπως ανταγωνιστική νομοθεσία, κρατικές ενισχύσεις, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα που θα ε, αφιερωθούν, ε, θα διοχετευτούν σε ιδιωτικά προγράμματα. Αυτά πράγματα θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένες ενέργειες και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα προγράμματα χρηματοδότηση μπορεί να ε, εκλειφθούν ως το πράσινο φως, εν λευκό επιταγή για κάποιες βιομηχανίες, οι οποίες θα αναπτύσσουν ε, δραστηριότητες σε αναπτυσσόμενες περιοχές του κόσμου, κάπου αλλού, πολύ μακριά. Αυτό που μας ανησυχεί επίσης είναι η ενεργειακή φτώχεια. Όπως ενδεχομένως θα γνωρίζετε, η Συνομοσπονδία των ε, Συνδικάτων ε, συμμετέχει στην πλατφόρμα ενέργειας. Η ενεργειακή φτώχεια εμάς μας απασχολεί πάρα πολύ. Όπως ξέρετε, το 10% των οικοκυριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν, δεν είναι σε θέση να θερμάνουν κανονικά τα σπίτια τους. Αυτό μας ανησυχεί πολύ και η στρατηγική μας είναι ότι τα κοινωνικά θέματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από συστήματα κοινωνικής προστασίας και ευημερία. Αυτό όμως είναι μία περίεργη απάντηση. Πρώτον, διότι έχουμε δει εδώ και πολλά χρόνια ότι οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένων των φόρων που καταβάλλονται από τα νοικοκυριά αυξάνονται συνεχώς. Και αν συγκρίνει κανείς αυτήν την τάση με την άλλη που αφορά στο διαθέσιμο εισόδημα, θα διαπιστώσει ότι οι δύο αυτές καμπύλες δεν εξελίσσονται παράλληλα. Επίσης, χάρη εκθέσεων όπως αυτή που δημοσίευσε η Μπρούγκελ τον Νοέμβρη ε, που πέρασε, ξέρουμε ότι οι πολιτικές για το κλίμα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών οδήγησαν ε, σε σημαντικές επιπτώσεις ως προς τον επιμερισμό που έχουν επηρεάσει πρώτα απ' όλα τα χαμηλά εισοδήματα τα φτωχά νοικοκυριά. Εξάλλου γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε και πολύ σημαντικές επενδύσεις για να μπορέσουμε να απομακρύνουμε τον άνθρακα από την ενωσιακή οικονομία. Υπάρχουν εξή σενάρια ότι θα έπρεπε να ε, εξαπλασιάσουμε τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποθήκευσης άνθρακα. Όμως στο έγγραφο αυτό δεν αναφέρεται το κόστος που θα προκύψει και πώς ακριβώς το κόστος αυτό θα επιμεριστεί στην οικονομία ανάμεσα στον ιδιωτικό τομέα και τα νοικοκυριά και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί σήμερα γνωρίζουμε στη Γαλλία, στο Βέλγιο, αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη. Εχθέ πήγα στην Πολωνία μαζί με τον συνάδελφό μου στην Κούρτικα και πρέπει να σα πω, τον κύριο Κούρτικα, και πρέπει να σα πω ότι μα απασχολεί πάρα πολύ η ενεργειακή φτώχεια. Πρέπει λοιπόν αυτά τα θέματα να αντιμετωπιστούν στη μακροχρόνια στρατηγική το να αμφισβητηθούν τα ωφέλη αλλά και το κόστος, πώς ακριβώς επιμερίζεται στην κοινωνία, αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος για να καθυστερήσει η απομάκρυνση του άνθρακα. Είναι πήγουσα. Αντίθετα, εγώ πιστεύω ότι το να προσέξουμε όλα αυτά τα θέματα κατ' ουσίαν σημαίνει ότι επιτρέπουμε την επιτάχυνση της ε, απομάκρυνης άνθρακα. Και όπως σας είπα, αν δεν προσέχουμε αυτά τα θέματα, θα έχουμε τελικά να κάνουμε με κοινωνικές αναταραχές. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι ε, θα πρέπει να ε, δουλέψουμε έγκαιρα για τους ε, επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού. Η στρατηγική να εφαρμοστεί με ένα τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να συμβαδίζει με την επιστήμη και να είναι κοινωνικά αποδεκτή και να μην προκαλεί αποκλεισμούς. Σας ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο σας εκ μέρους των συνδικάτων. Τώρα, κυρίες και κύριοι, προχωρούμε στον γύρο ερωτήσεων και απαντήσεων. Ήδη έχω σημειώσει ορισμένα ονόματα συναδέλφων. Πρώτος ο κύριος, ο Λίζε, μια στιγμή διακόπτη. Με συγχωρεί, μεταθέτει βέβαια τον κύριο Λίζε. Να επιτρέψουμε στον Επίτροπο να κάνει μια σύντομη τοποθέτηση. Διότι μετά θα χρειαστεί να αποχωρήσει. Πολύ σύντομα, λίγα σχόλια. Επειδή τέσσερα χρόνια τώρα ασχολούμαι με την κλιματική πολιτική και τη στρατηγική αυτή για δύο χρόνια. Ορισμένοι μιλούν για την ανάγκη φιλοδοξότερων στόχων, αλλά δεν έχει νόημα αυτό. Βλέπετε τα NDC στο Μητρό των Ηνωμένων Εθνών. Μπορεί να γίνει κάτι άλλο όμως. Να συγκριθούν οι χώρες που έχουν NDC, δηλαδή εθνικές δηλωμένες συμβολές και οι χώρες που έχουν εθνικούς σχεδιασμούς. Ούτε το ένα δέκατο από, αυτούς, από αυτές όμως τόσο δεν έχουν ανταποκριθεί. Λοιπόν, το να βάζετε υψηλότερους στόχους δεν έχει κανένα νόημα αν δεν υπάρχουν πολιτικές. Η διαφορά με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι εμείς έχουμε στόχους και όλες τις πολιτικές για την επίτευξη των στόχων. Και χάρη στην ε, φιλοδοξία εντό εισαγωγών του Κοινοβουλίου. Έχουμε και πιο φιλόδοξε πολιτικές. Άρα, η θέσπιση νέων στόχων σημαίνει και δημιουργία νέων πολιτικών. Και ακόμα δεν έχουμε αρχίσει να εφαρμόζουμε τι πολιτικέ που διαθέτουμε. Είναι δύσκολε να εφαρμοστούν, γιατί αν δείτε, έχουμε μειώσει τις εκπομπές μας από το 1990 στο 2017 κατά 22%. 0,8% τον χρόνο. Αυτή ήταν η ταχύτητα μειώση των εκπομπών. Τώρα έχουμε νομοθεσία που θα μας οδηγήσει το 2030 να, είμαστε, να διπλασιάσουμε το ποσοστό αυτό. Για την ώρα υπάρχουν πολλές χώρες μπέλη οι οποίες δεν εκπληρούν τους στόχους ανανεωσίμων και πολλές που δεν εκπληρούν τους στόχους ε, για την αποδοτική χρήση τη ενέργεια. Άρα μπορούμε να βάζουμε στόχους. Αλλά αυτό που χρειάζεται είναι να εφαρμοστούν οι φυστάμενε πολιτικές. Το να γίνουμε ουδέτεροι ως προς το κλίμα θα χρειαστεί βέβαια αύξηση των στόχων. Έχουμε ήδη ρήτρε αναθεώρησης για το 2023. Θα είμαστε λοιπόν ει θέση να αλλάξουμε τι πολιτικέ μα το 2023. Εμένα με ενισχύουν πιο πολύ οι πολιτικέ παρά οι αριθμοί. Είμαι πολύ πιο υπερήφανος που... Ε, μάλλον θα είμαι πολύ πιο υπερήφανος στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει φιλόδοξες πολιτικές και όχι φιλόδοξους στόχους. Η παρούσα στρατηγική ανοίγει τον δρόμο για φιλοδοξότερους στόχους εάν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ζητήσουν κλιματική ουδετερότητα. Θα έλθουν αυτά τότε. Δεύτερο, ρυθμισμένες τιμές στο σχεδιασμό αγοράς προσπαθήσαμε να ξεφορτωθούμε τις ρυθμιζόμενε τιμές όσο μπορούμε. Μόνο κατ' εξαίρεση για τα νοικοκυριά. Διότι θέλουμε ανταγωνισμό στι αγορές, ώστε η ενέργεια να γίνει φθηνότερη. Με ρυθμισμένες τιμές, άνωθεν δηλαδή, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Και επίση οι ρυθμισμένε τιμέ δεν στοχεύουν αυτού που τι χρειάζονται πραγματικά. Και αυτό στη στρατηγική μας λέμε, ας αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας. Ας φτιάξουμε κοινωνικές πολιτικές για να στηρίξουμε αυτούς που έχουν ανάγκη. Να έχουν δηλαδή ενεργειακά αποδοτικά σπίτια, να έχουν την υποστήριξη που χρειάζονται. Γιατί είναι καλύτερα να έχουμε πολιτική ρυθμισμένο τιμών από το να έχουμε κοινωνικές πολιτικές. Η τρίτη παρατήρηση και τελευταία είναι θα ήθελα η στρατηγική αυτή να γίνει κυρίαρχο στοιχείο στις συζητήσει για τις ευρωεκλογέ. Ο κόσμος δηλαδή να συζητήσει το επίπεδο φιλοδοξίας, την ταχύτητα αύξησης των στόχων και να δούμε όλα τα πολιτικά κόμματα να θέτουν το θέμα επιτάπητο. Αν ρωτήσετε τον κόσμο αν η πολιτική του κλίματος είναι σημαντική, θα σα πούνε 9 στου 10 ναι. Αν ρωτήσετε αν είναι το πιο σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα θα σα πούνε μόνο το 30% ναι. Ε, συγγνώμη που χρειάστηκε να επανέλθω. Αυτά ήθελα να σα πω. Σα ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, λέει η πρόεδρος Βαλεάν, που σχολιάσατε τι διάφορε παρουσιάσει. Τώρα, α έρθουμε στου συναδέλφου. Και πρώτο ο κύριο Ελίζε. Ευχαριστώ κύριε, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Επιτροπό καθώ και τα άλλα μέλη του πάνελ. Εγώ χαίρομαι πολύ για το έγγραφο τη Κομισιόν και πραγματικά αποτελεί πρόκληση, είναι φιλόδοξο. Δεν μιλούμε για ουδετερότητα ανθρακό, αλλά για ουδετερότητα κλίματο, απέναντι στο κλίμα δηλαδή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ομιλεί για καθαρό κέρδο ενό εκατομμυρίου θέσεων απασχόληση όταν θα εφαρμοστεί η ουδετερότητα στο κλίμα. Και μαζί με άλλα σενάρια και συνεχή ε, ανάπτυξη. Τώρα φεύγει ο Επίτροπο, είναι όμω άλλοι παρόντε από του εκπροσώπου τη Κομισιόν, καθώ και οι πάνελιστ. Θα ήθελα να ακούσω από το πάνελ εάν ο αριθμό αυτό δεν αμφισβητείται. Γιατί έχω ακούσει στην πολιτική ομάδα να τίθεται και ερωτήσει, δηλαδή σε ποιου υπολογισμού βασίζεται. Οι πάνελιστ συμφωνούν με την ανάλυση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα εκατομμύριο δηλαδή πρόσθετε θέσει εργασία. Μήπω είναι λιγότερε, μήπω είναι ακόμη περισσότερες. Οι εμπειρογνώμονε τι ε, πιστεύουν σχετικά με τον υπολογισμό αυτόν. είναι παρόν ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορείτε παρακαλώ να προσέλθετε να καθίσετε εδώ στα έδρανα του Προεδρείου. Ευχαριστούμε κύριε Λίζε για τις ερωτήσεις σας. Ο κύριος Μπλάνκο Λόπες. Eh, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι, αντικειμενικά το λέω, ότι η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο ε, σε αυτή την ε, θητεία που σε λίγο ολοκληρώνεται, ε, πραγματικά κάλυψαν τις υποχρεώσεις τους και τις ε, έκαναν τους ε, συμβιβασμούς που έπρεπε έτσι ώστε να καταπολεμήσουν, μάλλον να αγωνιστούν κατά της κλιματικής αλλαγής. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή αυτή η στάση του, ε, η αντικομφορμιστική, όταν δηλαδή θέτουμε πολύ υψηλούς στόχους, γιατί αυτός ο αγώνας για το κλίμα πρέπει να είναι διαρκής, συνεχής, μέχρι ότου καταφέρουμε να επιτύχουμε αυτήν την ουδετερότητα στην οποία αναφέρθηκε ο Επίτροπος ε, και να ε, αφαιρέσουμε τον άνθρακα από την οικονομία μας. Τώρα, η οδηγία των, ε, των ανανεωσίμων. Εγώ είμαι εισηγητής για το θέμα. Αλλά και εγώ προσωπικά και όλοι οι συνάδελφοι που ασχολήθηκαν μαζί μου με το θέμα αναφερθήκαμε στους στόχους του 2030 ως ε, ελάχιστους στόχους. Ε, γι' αυτό ε, ζητήσαμε αναθεώρηση που μπορεί να ξεκινήσει το έτος 2023. Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε, μπορούμε να πάμε πιο πέρα, πιο μακριά και πέρα από αυτό που έλεγε ο εκπρόσωπος της Νομοσπονδίας Συνδικάτων, ενδεχομένως η εξέλιξη του κόστους ε, θα μας δώσει την δυνατότητα να πάμε ακόμα παραπέρα, όπως ε, είδαμε και με τη μείωση κόστους ε, για τη διείσδυση των ανανεωσίμων. Κάδαμε μεγάλη δουλειά, πολλή δουλειά και πρέπει να συνεχίσουμε. Προσπαθήσαμε να εισάγουμε αυτούς τους στόχους για την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδυας ως ένα στοιχείο ε, ε, θεμελιώδες έτσι ώστε σε αυτήν ε, την ελεύθερη από άνθρακα Ευρώπη να μην υπάρχουν πολίτες, άνδρες και γυναίκες που να μένουν πίσω και επίσης αυτή η αφαίρεση του άνθρακα να μην αποτελέσει κριτήριο κριτικής μεταχείρισης πολιτών. Ο κύριος Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στον κύριο Κούρτικα που ε, αποτέλεσε επιτυχία η προσπάθειά του για την COP23 ε, στην Κατόβιτσε. Τώρα, για την μακροπρόθεσμη στρατηγική, θα πρέπει αυτή να εφαρμόζεται σε ολόκληρο τον κόσμο και όχι μόνο σε εμά. Και νομίζω ότι αυτό επισημαίνεται και στο τελικό έγγραφο της Κατόβιτσε. Αλλά Μπορείτε ίσως να εξηγήσετε πώ και οι άλλοι θα υιοθετήσουν την ίδια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Άκουσα με ενδιαφέρον επίσης τον εκπρόσωπο τη ε, βιομηχανία που η θέση τη μου φάνηκε επικοδομητική. Ωστόσο, ασχολούμαστε πολύ με την Κίνα και κοιτούμε τι θα κάνουν. Κίνα 2025. Ε, αυτοί έχουν μια καθαρή βιομηχανική στρατηγική. Εγώ θα ήθελα λοιπόν ένα Made in Europe 2030 διότι χρειαζόμαστε πράγματι τεχνολογίες για τον χάλιβα, για τα χημικά, για το τσιμέντο. Ήδη μας έχουν πάρει οι Κινέζοι τα ε, φωτοβολταϊκά και τις μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Εμείς εισάγουμε τις τεχνολογίες αυτές τώρα από τους Κινέζους. Όταν όμως εσείς ομιλείτε ή μάλλον λέτε ότι οι Γενικές Διευθύνσεις Εμπορίου και ανταγωνισμού ή ε, γενικής διαβιομηχανίας να, είναι, να υπάγονται στη γενική διεύθυνση βιομηχανίας Ίσως μπορεί να απαντήσει ο πρόσωπο τη Κομισιόν. Πώ θα αλλάξουμε την πολιτική αυτή, γιατί χρειαζόμαστε βιομηχανική πολιτική η γενική διαβιομηχανιας να ειναι να υπαγονται στη γενικη διευθυνση βιομηχανία. ισως μπορει να απαντησει ο προσωπο τη κομισιον πω θα αλλαξουμε την πολιτικη αυτη γιατι χρειαζομαστε βιομηχανικη πολιτικη η οποια να ανοιγει το δρόμο προ τα εμπρό. Βλέπουμε και πολλέ διαμαρτυρίε. Και εν ώψη των διαμαρτυριών αυτών, καλώ κάνουν τα εργατικά συνδικάτα και μιλούν για την κοινωνική δικαιοσύνη διότι ναι μεν στρατηγική για το περιβάλλον, αλλά πρέπει να υπάρχει και στρατηγική υπέρ της κοινωνίας, γιατί οι φτωχοί τελικώς καλούνται να πληρώσουν το λογαριασμό, είτε είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, είτε να αγοράσουν καινούριο αυτοκίνητο, είτε να ανακαινήσουν το σπίτι τους. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια νέα στρατηγική που θα επιτρέψει μια εξισορρόπηση και αυτό βεβαίω είναι καθήκον των χωρών μελών, γιατί είναι ζήτημα κοινωνική πολιτική. Αλλά με κάποιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπιστεί, με συντονισμό ίσω από πλευρά τη Κομισιόν και, και ημών εδώ των Ευρωβουλευτών. Ελπίζω η ταξόνομη να μας διευκολύνει, δηλαδή να, έχουμε, ε, να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα νέο σύστημα χρηματοδότησης για την πράσινη οικονομία. Ευχαριστώ. Γκέρ Μπράντι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. δηλώνω ικανοποιημένος με το έγγραφο μακροπρόθυμη στρατηγικής της Κομισιόν. Αυτή η προστιθέμενη αξία του να γνωρίζουμε που θέλουμε να φτάσουμε το 2050 είναι ότι μπορεί κανείς να υπολογίσει μετά προς τα πίσω και να δει πώς θα κάνει τα βήματα ώστε να φτάσει στον επιθυμητό στόχο. Είναι σημαντικό αυτό, αλλά για να επανέλθουμε στο σήμερα, το 2019, βλέπει κανεί και πόσο δύσκολο είναι αυτό. Το 2017 αυξήθηκαν οι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε ακόμα τα νούμερα του 2018, αλλά θα με πλήξει ε, πραγματικά εάν δούμε ότι υπήρξε μείωση. Βλέπετε και η εγκατάλειψη ε, του άνθρακα στην ε, ε Γερμανία και αυτή θα χρειαστεί χρόνο. Βλέπω και στη δική μου χώρα, την Ολλανδία, πόσο δύσκολη είναι η υπόθεση του περιβάλλοντος και του κλίματος όταν απαιτείται να ε, μεταφραστεί σε συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνονται στην πράξη. Άκουσα προσεκτικά όλα τα μέλη του πάνελ. Άκουσα τον ε, Επίτροπο να μιλεί για ε, το ότι οι φιλοξότεροι στόχοι χρειάζονται κοινέ πολιτικές. Ο κ. Μένσινγκ και αυτό με βρίσκει σύμφωνο, ο οποίο Μένσινγκ μίλησε για την ανάγκη μεγάλων επενδύσεων σε μελλοντικέ υποδομέ και ο κ. Ντάνη για την ε, καινοτομία που είναι επίση απόλυτα αναγκαία. Ταυτόχρονα ρυθμίζουμε εμείς το χρηματοδοτικό τμήμα, δηλαδή το πι μέχρι το 2027. Συζητούμε και το εγκρίνουμε στη βάση φέτος. Αυτό σημαίνει ότι τα επόμενα 10 χρόνια αποφασίζουμε τώρα περίπου πώς θα ε, δαπανίσουμε αυτό το 1 εκατομμύριο ευρώ. Και η ερώτηση ε, θα πρέπει να είναι δεν πρέπει να επανεξετάσουμε τις προτάσεις του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου ε, υπό το πρίσμα της μακροπρόθεσμης πολιτικής για να δούμε αν πραγματικά ε, σέβονται το κλίμα. Διότι αν συνεχίσουμε να επενδύουμε σε στοιχεία τα οποία δεν είναι ασφαλή για το κλίμα, ε, τότε στην πραγματικότητα βάζουμε την εκλοποδία στον εαυτό μας. Αυτό είναι μια ερώτηση προς όλο το πάνελ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ριβαζή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που υπάρχει αυτή η μακροχρόνια στρατηγική. Γιατί ως συνεισηγήτρια για τη διακυβέρνηση της ενέργειας μαζί με τους συναδέλφους προσπαθήσαμε να είμαστε φιλόδοξοι όσον αφορά τους στόχους για τα ανανεώσιμα κτλ. Αλλά η διακυβέρνηση αφορά την υλοποίηση, δηλαδή πώς τα παιδιά, οι χώρες μέσω των διαφανών ε, ε, σχεδίων θα υλοποιήσουν ε, και θα επιτύχουν τους στόχους αυτούς είπαμε θα μπορούσαμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι σε επίπεδο ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το 2030 γιατί είχαμε πει τότε 40% εάν επιτύχουμε ε, το 32% για τις ανανεώσιμε θα φτάσουμε στο 45% και θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο 60% για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα όμως έχουμε τρεις λέξεις κλειδιά. Ε, συνοχή, ε, ευθύνη και φιλοδοξία ευθύνη. Γιατί αν δείτε πώς είναι οι νέοι που βρίσκονται στους δρόμους αυτή τη στιγμή για το κλίμα, διαμαρτύρονται για το κλίμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, αυτή η Γκρέτα Τένμπερκ, η κοπελίτσα αυτή η μικρή, ε, η οποία οδήγησε όλους τους νέους ε, των ηλικίων να αρχίσουν να φωνάζουν για το κλίμα. Ε, αυτό πρέπει να είναι ο πρώτο στόχο για το κλίμα. Επίση, φιλοδοξία σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μπορούσε να είναι πιο μεγάλη. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, θα προσπαθήσουμε να ε, ε, ε, υπάρξουν επενδυτικά προγράμματα. Εσείς αναφέρεστε σε καινοτομία, αλλά η καινοτομία θα πρέπει να καλύψει αυτό το έλλειμμα του 3%. Θα πρέπει επομένως να βγάλουμε τις βιώσιμες υποδομές από αυτό το 3% του ελλείμματος, γιατί διαφορετικά δεν θα τα καταφέρουμε. Και επίση από πολιτικής απόψεως, αν θέλουμε ελεύθερες συναλλαγέ μεταξύ των χωρών, άρα θα γίνουν πιο πολλέ οι μετακινήσεις, ε, εισαγωγέ, εξαγωγέ. Μιλάτε, αναφέρεστε στη βιομηχανία, λέτε ότι η βιομηχανία θα πρέπει να ξαναέρθει στην ε, Ευρώπη, αλλά θα πρέπει να ξαναδούμε λίγο και αυτή τη φιλελεύθερη πολιτική μας, γιατί αύξηση συναλλαγών σημαίνει αύξηση μετακινήσεων. Επίσης, εάν ε, επενδύουμε στα ε, καύσιμα τα ορυκτά, δεν θα έχουμε καλό αποτέλεσμα. Εάν δεν αμφισβητήσουμε την ΚΑΠ έτσι όπως έχει καθοριστεί ε, σε σχέση με τη γεωργία, δηλαδή έτσι όπως την έχουμε συνηθίσει, δεν θα έχουμε καλό αντίκτυπο στο περιβάλλον και όσον αφορά τους βιομηχάνους. Μα η βιομηχανία θα πρέπει να ε, βγάλει αυτοκίνητα με ε, εκπομπές μηδενικές. Θα πρέπει να είμαστε συνεκτικοί. Έρχομαι στη συνοχή λοιπόν. Πρέπει να είμαστε λογικοί στις πολιτικές μας και στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Ευχαριστώ. Έχει, είχατε ένα λεπτό στη διάθεσή σας, πολύ ωραία τα λέτε και ήθελα να συνεχίσω να σας ακούω, αλλά ας προσπαθήσουμε να εστιάσουμε και να, μην κάνουμε σχόλια, να κάνουμε ερωτήσεις, να υποβάλουμε ερωτήσεις στους πανελίστες. Η συζήτηση επί, της, ε, ε, επί του ψηφίσματος ε, θα λάβει χώρα αργότερα. Η κυρία Νταλή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να πω ότι η στρατηγική της Κομισιόν μου φαίνεται πολύ θετική ε, και αυτός ο στόχος ε, για ε, μηδενικό και σε εκπομπέ άνθρακα. Μου φαίνεται πολύ κακό. Αλλά βεβαίω για το σκοπό αυτό θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν οι πάντε και τα πάντα. Στρατηγικέ, πολίτε, πολιτικοί κτλ. Έτσι ώστε και θα πρέπει ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε ε, και την κοινωνική ε, ισοτιμία και δικαιοσύνη. Ο Επίτροπο έλεγε προηγουμένω ότι είναι απαραίτητη ε, οπωσδήποτε η δέσμευση και η αποθήκευση του άνθρακα Πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως βλέπει τις τεχνολογίες ε, και πόσο γρήγορα θα μπορούσαν αυτές οι νέες ε, ε, στρατηγικές να εφαρμοστούν. Για τον κύριο Κούρτικα έχω να πω το εξής. Ως πρόεδρος της COP24 ξέρετε περισσότερα από μένα πώς φέρονται οι χώρες όταν κάνουν πολιτικές, όταν μιλάνε για το κλίμα και όταν τελικά κάνουν νομοθεσίες εσείς ε, σαν πρόεδρος της COP24 Κατοβίτσε ε, πώς μπορείτε να προωθήσετε την ε, πρόοδο ας πούμε και να, έτσι ώστε να αναλυφθεί δράση και πώς θεωρείτε ότι θα μπορούσατε να σπρώξετε λίγο τις ε, χώρες, ε, τους πολιτικούς, την κοινωνία των πολιτών, τη βιομηχανία, έτσι ώστε να επιτεχύνουν την προσπάθειά τους για να αντιδράσουν σε αυτά τα προβλήματα. Ε, επίσης, η δημιουργία του Ταμείου ε, Δίκαιης ε, Μετάβασης. Ε, πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ καλό που έρχεστε εδώ σαν εκπρόσωπο συνδικάτων και μας λέτε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε νέα τρόπο αντίδρασης. Ναι, αλλά πώς θα τα διαπραγματευτείτε αυτά και πώς σε αυτήν την μετάβαση και τη μεταβατική περίοδο θα καταφέρετε να φέρετε μαζί σας στην προσπάθεια αυτή όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ελπίζω οι απαντήσεις ε, να είναι πιο σύντομες. Ο κύριος Άικαουτ. Έχετε κάτι καινούργιο να προσθέσετε? Δεν θα σας ε, απογοητεύσω. Έχω τρεις πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Η μία είναι προς τον κύριο Πετριτσόνη, η μία προς τον κύριο Τσχα και η μία προς τον κύριο Μέντσινγκ πρώτη στην την Επιτροπή τον κύριο Πετριτσόνε. Ξέρετε ότι έχουμε κάνει πολλέ συζητήσει και εσεί συνεχίζετε να λέτε ότι το μείον 40% είναι πάρα πολύ καλό για το Παρίσι. Διαφωνούμε ριζικά, αλλά ε, μία ερώτηση για να μου εξηγήσετε λιγάκι το δικό σα το πρότυπο. Το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε για να φτάσουμε στο μείον 8 μέχρι το 2050, μείον 40 στο 2030. Αυτό ε, είναι ακριβώ η λύση για να είμαστε αποτελεσματικοί ως προς το κόστος. Όμως έχουν μειωθεί παραδείγματος χάνει τιμές ε, των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας. Άρα και για το μείον 80 θα μπορούσε κανείς να πει ότι πρέπει να προχωρήσουμε και μπορούμε πιο γρήγορα, αλλά η Κομισιόν λέει ουδέτερη μόνο το 2050. Άρα δηλαδή το μείον 40 που συμφωνήσαμε το 2011 και εγκρίθηκε το 2014, ένα χρόνο πριν από το Παρίσι, ποιο είναι αυτό το μοντέλο σας που με το μείον 40 είμαστε στο σωστό δρόμο ε, και ε, δεν δέχεστε ότι αυτό είναι χάσιμο χρόνο. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Μετά στον κύριο Κούτσκα, όταν θα πάμε το Σεπτέμβριο στο Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ, τι απάντηση θα του δώσετε, γιατί εκείνο ζητάει περισσότερο φιλόδοξα προγράμματα. Και ποια θα είναι η απάντηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι σε 9 Μαΐου συζητήσαμε μια, ένα πολύ καλό χάρτη πορεία και ήταν μια πολύ χαρούμενη και ωραία συζήτηση. Αυτά θα πείτε στο Γενικό Γραμματέα και προς τον κύριο Μένσινγκ. Άκουσα ο, τη βιομηχανική σας ατζέντα ε, και θα μπορούσαμε ίσως ε, να συμφωνήσουμε γιατί πράγματι πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα αλλά κάπου ζητάτε ε, ρυθμιστικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, περισσότερα χρήματα για τη βιομηχανία, πολλά που θέλει η βιομηχανία αλλά όλα αυτά καταλήγουν στο χρήμα. Και σας ερωτώ, εσείς ανταυτού τι θα μας δώσετε. Δηλαδή θα συμφωνήσετε ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο τίμημα για τον για τον άνθρακα ή θα πληρώσουν τελικά οι πολίτες. Σας απασχολεί λιγάκι ο δίκαιος επιμερισμός ε, και για τη βιομηχανία. Δηλαδή ε, να λέτε ότι εντάξει τότε θα πληρώνουμε περισσότερο για τον άνθρακα, για τη μη ταξική στρατηγική στην Ευρώπη, γιατί αυτά θέλουμε να ακούσουμε. Ε, δεν μπορεί κανείς να ζητάει πράγματα και να μην δίνει τίποτα. Ελπίζω, κύριε Πρόεδρε, αυτά να μην τα είχατε ξανακούσει, να ήταν νέα. Το θέμα δεν είναι αν ήταν νέα καινούργια ή όχι, αλλά ε, δεν ε, το χρόνο. Ναι, αλλά και εγώ δεν μπορούσα και να είμαι και ε, να πω κάτι καινούριο και να κρατήσω και το χρόνο. Ε, δεν γίνεται, δεν γινόταν αυτό. Μην ξεχνάτε όμως ότι ακολουθούν εκλογές. Πρέπει να κάνουμε και μια προπόνηση για τις ομιλίες. Και μην ξεχνάτε, ο Επίτροπος είπε ότι θα πρέπει τη συζήτηση να την κρατάμε ενδιαφέρουσα και για τους πολίτες. Η κυρία Γκούντελαντ, ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους ομιλητές ως ε, συνεισηγήτρια της Σοσιαλδημοκρατικής Ομάδας για το LTS. Χαίρομαι που έγινε αυτή η συζήτηση και χαίρομαι ε, που ε, Συμφωνώ και εγώ, όπως είπε και η Επιτροπή, υπάρχουν πολλές καλές προτάσεις ε, που εντάσσονται σε αυτή τη στρατηγική. Θέλω όμως να πω στην Κομισιόν ότι εμένα αυτό που με απασχολεί είναι ότι δεν προσφέρεται αυστηρούς στόχους για το 2030 και αυτό είναι λάθος. Να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί είναι τόσο επιφυλακτική στο θέμα αυτό. Γιατί πιστεύω ότι θα ήταν ε, πιο προβλέψιμο για τη βιομηχανία το να μπορούμε να δείξουμε ε, ποιο δρόμο θα ακολουθήσουμε έτσι ώστε να μην καθυστερήσουμε και να μην έχουμε πολλές δυσκολίες για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Επίσης υπάρχει και κάτι άλλο. Εγώ δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαφωνεί με όλα αυτά. Νομίζω συμβαίνει το αντίθετο. Πιστεύω όμως ότι φοβόσαστε το Συμβούλιο και αυτό είναι το πρόβλημα. Ε, γιατί λέτε τώρα και επιχειρηματολογείτε σαν να μην θέλετε να ε, βελτιώσετε τους στόχους για το 2030. Είναι σαν να μην θέλετε να μας βοηθήσετε. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κουρτσίκα για την ε, πολύ καλή COP24, πολύ καλή οργάνωση, είχατε ένα πολύ σημαντικό ρόλο και επίσης και ε, το εγχειρίδιο με τους κανόνες ήταν πάρα πολύ καλό, αλλά οι φιλοδοξίες είναι σημαντικές για το μέλλον. Και θέλω να ακούσω τις απόψεις σας για το πώς θα μπορούσαμε να σκίσουμε περισσότερη πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να είναι πιο φιλόδοξη ως προς το μέλλον. Η κυρία Μέτς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σωστή η ιδέα μακροπρόθεσμη στρατηγική. Θα είμαι σύντομη. Πολύ σωστά είπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι, αν και μακρηγόρησαν λίγο. Διερωτώ με, στα οχτώ σενάρια που παρουσιάζεται και κυρίω απευθύνω το ερώτημα στην Κομισιόν, όλα περιλαμβάνουν και την πυρηνική ενέργεια σε τουλάχιστον 10%. Ούτε ένα σενάριο δεν υπάρχει 100% ε, ανανεώσιμε ενέργειες. Καμία επιλογή χωρί πυρηνικά χωρίς πυρηνικά εργοστάσια δηλαδή, και νομίζω ότι είναι βαρύ σφάλμα να μην λαμβάνετε λαμβάνεται υπόψη και μια επιλογή χωρίς πυρηνική ενέργεια. Γιατί αυτό. Τουλάχιστον να προβλέψετε μια επιλογή χωρίς πυρηνική ενέργεια. Δεν χρειάζεται βέβαια να εξηγήσω ποιε είναι οι αρνητικές επιπτώσεις της πυρηνικής ενέργειας. Ευχαριστώ κυρία Μέτς. Πραγματικά ε, σύντομότατη. Ο κύριος Ντάνς, ευχαριστώ πολύ σύντομα. Σωστή η προσέγγιση της Κομισιόν. Ορισμένοι εξημών ίσως και να μην συμμετάσχουμε στις ευρωεκλογές του Μαΐου. Ε, λέω ίσως. Το πρόβλημα που βλέπω πάντοτε είναι ότι οι εγχώριες συζητήσεις και πολιτικές που θα διεξαχθούν στις χώρε μέλη μας δηλαδή, είναι πάρα πολύ διαφορετικές από τη συζήτηση που διεξάγεται σήμερα εδώ. Ο κ. Κούρτικα, για τον κ. Κούρτικα, δηλαδή, πήγαμε στο, σε, στο ΣΕΙΜ στην Πολωνική Βουλή δηλαδή και αυτά που ακούσαμε είναι ότι ποτέ δεν θα πάρετε τον ανθρακά μας, ποτέ δεν θα μας στερήσετε τον ανθρακά μας δηλαδή. Βάζω εδώ την Πολωνία επειδή τυχαίνει να είστε εσεί εδώ. Αλλά αυτά συμβαίνουν παρόμοια πράγματα σε κάθε χώρα μέλο. Πώ θα γεφυρώσουμε την, ε, ε, το κενό αυτό, την απόσταση αυτή. Να συμφιλειώσουμε δηλαδή του Ευρωπαίου πολίτε που είπατε ότι είναι απόσπαστο μέρο, είναι αλήθεια. Από την άλλη μεριά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε και λαϊκιστέ οι οποίοι ευχαρίστω εκμεταλλεύονται του φόβου των ανθρώπων. Χρειάζονται ε, να δαπανηθούν χρήματα και να αναλυφθεί η δράση, αλλά εκτό από αυτό χρειαζόμαστε και μια πολιτική στήριξη Έχετε καμιά ιδέα και καμιά συμβουλή για όσου εξημών ε, θα κατέβουμε στις ευρωεκλογέ. Σα ευχαριστώ όλες και όλου, λέει η πρόεδρος Βαλιάν. Αγαπητοί ε, προσκεκλημένοι, πολλέ ερωτήσεις ε, και ορισμένες μάλιστα πραγματικά περίπλοκες. Θα χρειαστεί, έχουμε κι άλλο πανελ μάλλον, αλλά θα χρειαστεί να είστε σύντομοι στι απαντήσεις σα. ίσως να συνοψίσετε και όλα σε ορισμένες απαντήσεις. Θα σας παρακαλέσω να μην μιλήσετε πάνω από πέντε λεπτά. Ας αρχίσουμε τον κύριο Κούρτικα. Χα, χα. Ε, πραγματικά είναι περίπλοκο το καθήκον που μου αναθέτεται. Ωστόσο η συζήτηση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας και ιδίω για αυτό το trade-off, αυτό, αυτή την ανταλλαγή, το παζάρεμα, αν είναι νέο ή αν είναι επίκαιρο, είπε ο κ. Σέικχαουτ. Αυτή είναι η ερώτηση που απασχολεί και την κλιματική μας πολιτική. Αν θέλουμε κάτι το νέο, χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Αν θέλουμε να είμαστε σύντομοι, θα πρέπει να παραμείνουμε στα παλιά και γνωστά. Υπό την έννοια αυτή θα είναι αρκετά περίπλοκο να βρούμε νέες, ερω... απαντήσεις αν δεν δώσουμε σε αυτούς επαρκή χρόνο για προβληματισμό, να δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε και μέχρι πού μπορούν να μας ακολουθήσουν οι κοινωνίες μας. Λέχθηκε και ευχαριστώ την κυρία Ριβασί που μίλησε για ζητήματα ευθύνης, συνοχής κλπ η οποία επέμεινε πολύ στο θέμα της ευθύνη και νομίζω ότι έχει δίκιο. Πάντως αυτό που παρατηρώ, ίσως βέβαια μόνο ε, στους δρόμους της Δυτικής Ευρώπης και λιγότερο ε, στην Ανατολική Ευρώπη, δηλαδή έχουμε και τα δύο ε, έχουμε ανθρώπους που κατεβαίνουν με τα κίτρινα γυλαίκα και άλλους που πηγαίνουν στις διαδηλώσεις υπέρ του κλίματος. Πώς θα γεφυρώσει κανείς τις πολιτικές αυτές οπτικές για τις βιομηχανικές πολιτικές, πολιτικές ε, για το κλίμα και πολιτικές εν τέλει υπέρ της κοινωνίας. Αυτά θα κρυθούν βέβαια και στις ευρωεκλογέ που θα γίνουν φέτος. Ασφαλώς και θα είναι ε, δύσκολη και περίπλοκη η πρόκληση. Πολύ εξημών και σας ευχαριστώ ε, κύριε Ελίζε, Λάινεν, Μπλάνκο Λόπεθ, κυρία Ντάλι. Πολύ λοιπόν από εσά μιλήσατε για την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η δίκαιη μετάβαση. Αυτό που αντιμετωπίζουμε όλο και περισσότερο δεν είναι μόνο οι επιπτώσεις που διαπιστώνουμε ας πούμε σε βιομηχανικές περιοχές όπως της Σιλεσίας για παράδειγμα που γνωρίζετε ότι είναι βιομηχανική περιοχή και υπάρχει ανάγκη να ενισχύσουμε τον κόσμο εκεί να μετακινηθούν από τις βιομηχανικές δουλειές που κατέχουν σήμερα σε άλλες δουλειές στο μέλλον. Αυτό είναι μια από τις πτυχές της δίκαιης μετάβασης. Άλλη που έχει σχέση με τις παλαιές, και έχει σχέση μάλλον με τις παλαιές βιομηχανίες. Πιο σημαντικό ωστόσο είναι το ερώτημα της συνολικής ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Και τα είπε αυτά και η βιομηχανία. Τι είδους δηλαδή καινοτομία θα χρειαστεί σε μια κοινωνία ουδέτερη απέναντι στο κλίμα και καθοδόν προς αυτήν, γιατί αυτός είναι και ο στόχος. Τι μπορεί να βοηθήσει, τι μπορεί να συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμβαίνουν πολλά. Εκεί δηλαδή κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αν δείτε όμως τι γίνεται με τη βιομηχανία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πέντε από τους έξι μεγαλύτερους παραγωγούς φωτοβολταϊκών είναι στην Κίνα. Το ίδιο ε, η παραγωγή ανεμογεννητριών, μπαταρίες, ε, μπαταρίες για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ηλεκτρικά λεωφορεία. Όλα αυτά ε, είναι στην Κίνα, προέρχονται από την Κίνα. Πρέπει να το λάβουμε λοιπόν αυτό στην σκέψη μας για μια στρατηγική που θα πρέπει να βασίζεται και σε ένα κοινωνικό πυλώνα και σε ένα πυλώνα για το κλίμα και στόχους βέβαια αναλόγως. Και αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι πρέπει να το ε, παρουσιάσουμε στους πολίτες ως όραμα μιας κοινωνίας, δηλαδή πώς θα διαμορφωθεί η κοινωνία του δεύτερου μισού του 21ου αιώνα. Γιατί αν κολλήσουμε στις συζητήσεις περί κόστους, αν κολλήσουμε στις συζητήσεις περί των αυξανόμενων τιμολογίων που ε, ε, λαμβάνουν οι πολίτες του λογαριασμού του δηλαδή για, λόγω αυξημένου κόστους ενέργειας, τότε χάνουμε το στόχο. Γιατί δεν τα καταφέρνουμε να δώσουμε στον κόσμο ένα θετικό όραμα μιας κοινωνίας που θα είναι ουδέτερη για το κλίμα, η δράση της δηλαδή. Και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε την ποιότητα ζωή των πολιτών όπω την βλέπουν οι ίδιοι. Αυτή η συζήτηση μένει να γίνει ακόμη και δεν είναι εύκολη. Νομίζω πάντως ότι είναι και αναγκαία. Και η δίκαιη μετάβαση βέβαια δεν αφορά μόνο την κοινωνική πολιτική, αφορά και την βιομηχανική πολιτική και το συντέριασμα των δυο, καθώς και περιφερειακή πολιτική, γιατί όταν μιλούμε για ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας, το ζήτημα είναι, ναι, μπορούμε να συζητήσουμε τα νούμερα. Δεν είμαι σε θέση ε, να συζητήσω τα νούμερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόβαλε το αναριθμό αυτό μπορεί να το εξετάσει πάλι. Αν πάντω αυτό το 1 εκατομμύριο νέων θέσεων εργασία όντω δημιουργηθούν, το ερωτηματικό είναι ποια θα είναι η περιφερειακή κατανομή αυτών των θέσεων εργασίας. Πού δηλαδή θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, πού εργασία, που δηλαδη θα δημιουργηθουν θέσει εργασια που θα χαθουν θεσει εργασία. και αυτο μα φερνει σε αυτο που ειπε η κυρία Ντάλη για ένα ταμείο δίκαιης μετάβαση. Είναι σημαντικό να το κρατήσουμε αυτό, να το έχουμε υπόψη μα, για να μπορέσουν να πάνε να κινηθούν παράλληλα οι δύο διαστάσεις. Δεν μπόρεσα να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, διότι αυτό θα σήμαινε μια πραγματικά πληρέστατη συζήτηση. Πάντως είμαι υπερήφανος για το αποτέλεσμα της COP24. Χαίρομαι πολύ που εμείς ήμασταν οι οικοδεσπότες της ε, διάσκεψης Κατόβιτσε και μπορέσαμε ομόφωνα να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για το ποιοι θα είναι οι κανόνες για την κλιματική πολιτική του μέλλοντος. Και αυτό δημιουργεί ένα πλαίσιο μέσα σε ένα πενταετή κύκλο που θα πρέπει να ε, δίνουμε απαντήσεις στις ερωτήσεις που δημιουργούνται. Και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για όλους, προς όλους. Και αυτό είναι η σημαντική συμβολή της Κατόβιτσε στην ε, συζήτηση που διεξάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρος Βαλεάν. Ο κύριος Μέσνικ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομο όσον αφορά το θέμα του ενός εκατομμυρίου θέσεων. Δεν μπορώ να κάνω υπολογισμό. Νομίζω οι περισσότερες θέσεις τα τελευταία χρόνια ήταν στις ε, Βρυξέλλες, αλλά αυτό το λαμβάνουμε υπόψη μας στους υπολογισμού μας. Ε, Ευρώπη 2030 βλέπετε ότι και εμάς μας απασχολεί αυτό. Αν περάσουμε μέσα από αυτή τη μεταβατική περίοδο, νομίζω ότι ε, το να έχουμε το Made in Europe. Αυτό είναι και η πρακτική που ακολουθούν και οι Κινέζοι, οι Αμερικανοί. Εμείς ε, δεν έχουμε τον πληθυσμό να αυξάνεται τόσο πολύ όσο στην Κίνα και την Αμερική. Γι' αυτό ε, ζητάμε και μεγαλύτερες επενδύσεις. Και χαίρομαι να απαντήσω στην τρίτη ερώτηση του κ. Άκχαουτ, με τον οποίο γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό. Θα επενδύσουμε, θα κάνουμε μεγάλες επενδύσεις για στήσει οποιοδήποτε ε, σύστημα στήριξη ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 20% είναι από το κράτος και το 80% είναι από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ε, και αυτό είναι ένα ένιγμα που πρέπει να το λύσουμε. Έχουμε εργαλείο όπως το Spire. Δεύτερον, εάν θέλουμε να ε, διπλασιάσουμε την κατανάλωση ενέργειας στην Ευρώπη, πώς μπορούμε να το κάνουμε χωρίς να αυξήσουμε τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους πολίτες και για τις βιομηχανίες. Αυτό είναι ένα δύσκολο ερώτημα που πρέπει να ε, απαντήσουμε. Ακόμα το ένιγμα δεν έχει λυθεί. Εκεί λοιπόν βρισκόμαστε, αρχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, έχουμε άλλα 10 χρόνια, όμως ε, τα ανοίγματα που πρέπει να λυθούν κρατημέλη και ακομισιών είναι τεράστια. Όσον αφορά το CCS, ε, δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, ερώτηση κυρία Ντάλη, πιστεύω ότι πλέον φτάνουμε σε ένα επίπεδο όπου έχουμε ξεπεράσει το να λέμε αυτή η α ή τεχνολογία είναι κατάλληλη. Χρειαζόμαστε το CCS ε, κοντά στη βόρεια ε, θάλασσα. Εκεί υπάρχουν ε, εγκαταστάσεις, όχι στο κέντρο της Ευρώπης, σε το υδρογόνο αλλού, αλλού ο άνθρακας. Βλέπετε όμως ε, ότι λαμβάνουμε όψη μας τις εκπομπές που δεν μπορούμε να απομακρύνουμε με άλλο τρόπο. Και τέλος, μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για πλήρη ανασυγκρότηση της βιομηχανίας στην Ευρώπη. Δεν είναι απλά ένας νέος χώρος και νέα εγκατάσταση. Μέχρι σήμερα οτιδήποτε από αυτά που βλέπετε δεν θα υπάρχει μέχρι το 2050. Και ε, να πω και κάτι, με βάση αυτά που, είπαν, που είπε ο Πολωνός συνάδελφος, ε, το υδρογόνο να κατασκευάζεται στην Πολωνία και να μεταφέρεται εδώ, αυτό δεν το θέλουμε. Η λογική του να έχουμε ενιαία βιομηχανία είναι ότι θα συνδέονται ε, τομεί που παλαιότερα δεν συνδέοντουσαν. Υποτιμάτε, λέτε, σε εμά την πρόκληση, αλλά δεν το κάνουμε αυτό. Και γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε αυτές τις ε, τεράστιες επενδύσεις στην Ευρώπη. Δεν σας ζητάμε να πληρώσετε, απλά σας θέλουμε να μας βοηθήσετε στις συζητήσεις ε, για επενδύσεις με τις τοπικές εταιρείες. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν πρέπει να μετακυλήσουμε το κόστος ε, στην κοινωνία ή στους πολίτες. Ορισμένες από τις απαντήσεις, κύριε Άικχαουτ, δεν τις έχουμε αυτή τη στιγμή. Είναι τεράστια τα προβλήματα, αλλά βλέπετε ότι οι επενδύσεις πρέπει να έρθουν από εμά και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε λύσεις για αυτά που εισάγουμε στην Ευρώπη. Γιατί τελικά δεν είμαστε μικροί με 500 εκατομμύρια καταναλωτές, αλλά θα είμαστε τελείως διαφορετικοί σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο, πιο καταρκεμασμένοι από ποτέ. Και το σύστημα σέρφικ είναι μέχρι τον Απρίλιο μαιο θα έχουμε τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική μας. Ε, προσπαθούμε να βρούμε τις απαντήσεις Είμαστε επεπισμένοι, Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με 10-20 μεγάλα πιλωτικά προγράμματα για να μπορέσουμε να αποδείξουμε στη βιομηχανία ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αν δεν αρχίσουμε να κάνουμε το πρώτο βήμα, τότε ε, δεν νομίζω ότι θα προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε θα απαντήσω στα γαλλικά, μια και είναι η μητρική μου γλώσσα. Όσον αφορά την απασχόληση, δεν κάνουμε μοντελοποίηση οικονομετρική ε, γι' αυτό δεν είμαι σε θέση να απαντήσω στην ερώτηση ε, ε, περί του ενός εκατομμυρίου θέσεων εργασίας. Όμως, και λόγω των συχνών επαφών που έχουμε με τα μέλη μας σε όλους τους τομείς και σε όλη την Ευρώπη, αυτό που ξέρουμε λέω, είναι ότι οι τομείς αυτοί οι οποίοι υποτίθεται θα πρέπει να προωθήσουν την τεχνολογία χαμηλής, χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ε, είναι αυτοί που έχουν ε, την τάση να οδηγούνται ε, σε ε, ψηφιοποίηση, αυτοματοποίηση, ε, αλλαγή έδρας ε, και επομένως μείωση των θέσεων εργασίας. Πάντως, η αύξηση των θέσεων εργασίας θα πρέπει να βασιστεί, να στηριχτεί και στο γενικότερο μακροοικονομικό και βιομηχανικό πλαίσιο, γιατί το δυναμικό των θέσεων εργασίας δεν αφορά μονάχα την τεχνολογία, αλλά επηρεάζεται και από το οικονομικό μοντέλο. Ε, ξέρουμε ότι τα φωτοβολταϊκά ας πούμε αποτέλεσαν καταστροφή ε, για τη βιομηχανική απασχόληση στην Ευρώπη, όμως ακούμε θετικά μηνύματα για τις ανεμογεννήτριες ε, και για ανανεώσιμες Ξέρουμε ότι είναι πολλές πάντως οι βιομηχανίες οι οποίες αναγκάζονται να φύγουν από την Ευρώπη γιατί γιατί ε, ακόμα και ε, υπάρχουν βιομήχανοι που μας λένε ότι είναι πολύ πιο φτηνό ε, να κάνουν ακόμα και τους πύργους, τα πόδια τέλο πάντων των ανεμογεννητριών να τα κατασκευάζουν στην Κίνα και να τα φέρνουν εδώ με, το, με τα μεταφορικά και παρόλα αυτά κοστίζει φτηνότερα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει και μια τεράστια προσπάθεια για τη μείωση των εκπομπών στις διεθνείς χερσαίες μεταφορές. Αυτό είναι απολύτως απολύτως απαραίτητο γιατί οπωσδήποτε ε, συμβάλλει πολύ στο πρόβλημα. Ε, κατανοώ ε, τα όσα είπε η κυρία Νταλή και ευχαριστούμε βεβαίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξη που έδωσε στις προτάσεις μας να δημιουργηθεί ένα ταμείο δίκαιης μετάβασης το εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο, όχι από το Συμβούλιο. Ε, η πρόταση που έγινε λοιπόν ε, για την δημιουργία ενός ταμείου 4,8 δις ε, για το επόμενο πι δελτα είναι πολύ καλό, είναι θετικό, ωστόσο πρέπει να προσέξουμε. Αυτό που μας ζητούν οι ε, εργαζόμενοι, των οποίων η θέση επηρεάζεται από την μείωση του ε, άνθρακα, είναι οπωσδήποτε κοινωνική προστασία και ενδεχομένως ανακύκλωση και ε, άλλη ε, και, και μετεκπαίδευση κτλ. Ε, αλλά αυτό που μας ζητούν κυρίως είναι ε, να δοθεί μια νέα πνοή στις περιοχές αυτές οι οποίες θα έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο από την μείωση του άνθρακα στην νότια ας πούμε Πολωνία όταν πηγαίνουμε ε, στις ε, ε, λεκάνες άνθρακα της Βουλγαρίας και μιλάμε με τους εργαζόμενους στον τομέα, ναι βεβαίως κατανοούν ότι θα πρέπει η οικονομία να απελευθερωθεί από τον άνθρακα, αλλά εάν κλείσετε το ορυχείο μου, εάν κλείσετε την, το θερμοηλεκτρικό σταθμό μου, τι θα κάνω, κάτι θα πρέπει να κάνω. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να προλάβουμε να προβλέψουμε. Χωρίς σωστή βιομηχανική ε, πολιτική κάποιοι εργαζόμενοι, κάποιοι πολίτες της Ευρώπης θα αντιμετωπίσουν εξαιρετικά μεγάλα και πολλά προγράμματα, προβλήματα. Επίσης, η ποιότητα των θέσεων εργασίας είναι αμφισβητήσιμη. Ε, μιλάμε βέβαια και για κάποιους τομείς όπου ιστορικά τα συνδικάτα έχουν δύναμη, μπόρεσαν να διαπραγματευτούν συλλογικές συμβάσεις με αξιοπρεπείς όρους εργασίας και μας ζητούν να εγκαταλείψουμε τους τομείς αυτούς. Ε, υπάρχουν όμως και άλλοι τομείς που δεν έχουν συλλογικές συμβάσεις, ε, οι συνθήκες εργασίας και αμοιβή είναι πάρα πολύ χειρότεροι από ό,τι στους παραδοσιακούς λεγόμενους τομείς. Επομένως θα πρέπει να σιγουρευτείτε ότι θα γίνει η μετάβαση, αλλά σιγουρευτείτε ότι θα ε, ε, υπάρχει και η απαραίτητη πρόβλεψη και ότι θα υπάρχει και η απαραίτητη ε, τροποποίηση της κοινωνικής ασφάλειας, της μέρημνας, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μην βρεθούν ξαφνικά χωρίς κανένα όπλο στα χέρια τους. Πολλές ερωτήσεις για την Κομισιόν. Τι έχετε να μας πείτε. Πρώτο, 2030 έναντι του 2050. Πολλοί θεωρούν ότι υιοθετεί κανείς μια πολιτική σήμερα, την, ε, την ε, εφαρμόζει γραμμικά και λύθει το πρόβλημα. Δεν συμβαίνουν έτσι τα πράγματα. Είχαμε τις τελευταίες δύο δεκαετίες μια πρόοδο, εγκρίναμε νομοθεσία που για τα επόμενα δέκα χρόνια ενισχύει την πολιτική αυτή σημαντικά και αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι ότι θα πρέπει να καταστεί ακόμα οξύτερη αυτή η πολιτική μέχρι το 2030. Ε, έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Εάν κάνετε, την προβολή σε, κάνετε γραμμική προβολή ε, δεν αποδίδει, δεν λειτουργεί. Αν δείτε τι γίνεται σε ό,τι αφορά την αύξηση του ΑΕΠ τα τελευταία 7 χρόνια, αυτά που αποφασίσαμε να κάνουμε στην Ομοθεσία για τα επόμενα 13 χρόνια, θα δείτε ποια θα είναι η πρόοδος της καμπύλης. Ορισμένες από τις πολιτικές για τις μιλούμε πρέπει να εφαρμοστούν και έχουμε και πολύ σημαντικά σημεία εχμής. Αν δεν λυθούν αυτά τα σημεία εχμής, ε, δεν είναι δυνατόν μια ε, γραμμική ε, πρόοδος να σας επιτρέψει να φτάσετε εκεί που επιθυμείτε. Αν εξετάσετε την αποδοτική χρήση της ΕΝΕΓΕ έχουμε στον, στην νομοθεσία ένα στόχο 32,2%. Δεν θα πετύχει όμως αν δεν λύσουμε το θέμα της, ε, του σημείου εχμής της χρηματοδότησης, διαθεσιμότητα της χρηματοδότησης. Πώς θα μεταφέρεται η χρηματοδότηση από τους μεγάλους θεσμούς στους μικροχρήστες. Αν αυτό το πρόβλημα μπορεί κανείς τότε ε, να κλιμακώσει προς τα πάνω την ε, πολιτική αυτή. Αν δεν λύσετε τα σημεία αυτά εχμής, δεν τα, διαλύσετε τα σημεία αυτά εχμής, δεν θα επιτύχετε τίποτα. Με όλες τις επιπτώσεις και στην αποανθρακοποίηση αλλά και στην απασχόληση, γιατί μιλούμε και για ανακαινήσεις ε, κτηρίων τοπικά. Υπάρχει λοιπόν μια συνέχεια που δεν είναι όμως μαθηματική. Είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι πολιτικές το 2050 δεν αποτελεί σχέδιο δράσης. Δεν αποτελεί στρατηγική με την έννοια ότι να ειδού τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε. Να με συμπαθάτε, πάνω από 30 χρόνια υπηρετώ στο Ευρωπαϊκό Δημόσιο, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε σήμερα τι είδους νομοθεσία θα χρειαστούμε το 2040. Μπορούμε να πούμε όμως ποιες, ποιους στόχους θα πρέπει να επιτύχουμε το 2050 και να προχωρήσουμε με σταδιακή βελτίωση της ε, νομοθεσίας. Μου άρεσε αυτό που είπε ο κ. Γκερμπράντι. Βάζει κανείς ένα στόχο και μετά βαδίζει προς τα πίσω έτσι ώστε να δει τι είδους νομοθετικές συνθήκες χρειάζεται και πότε τις χρειάζεται. Και αυτό προσπαθούμε να προτείνουμε με τη στρατηγική και την στήριξή της. Και η στήριξη δεν μπορεί να γίνει μόνο στις Βρυξέλλες. Δεν θέλω να είμαι ανάγωγος προς το Κοινοβούλιο, αλλά δεν μπορεί να γίνει μόνο από το Συμβούλιο, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να φτάσει σε βάθος σε όλες τις χώρες μέλη, γιατί το ζήτημα παρά είναι μεγάλο για να κρυθεί στις Βρυξέλλες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την φύση της μετάβασης, μιλούμε για βιομηχανική πολιτική. Συμφωνώ με αυτό που είπατε πριν Made in China 2025. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο Made in Europe 2050. Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά θα χρειαστεί να μετατρέψουμε τη βιομηχανία μας έτσι ώστε να μην είναι μόνο απαλλαγμένη από άνθρακα, από υπομπές δηλαδή ε, ε, οξυδίων του άνθρακος, αλλά να είναι και ανταγωνιστική. Και για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξει η τρέχουσα οικονομική ε, δόμησή της για να παραμείνει ανταγωνιστική για τα επόμενα 30 χρόνια και να συνεχίσει να προσφέρει ευημερία στην Ευρώπη. Ωστόσο, έχω ακούσει τα τελευταία 30 χρόνια παράπονα από παντού, από το Κοινοβούλιο, από τα συνδικάτα, από τη βιομηχανία. Έχουμε πράγματι μια εύθραυστη οικονομική κατάσταση. Τα καταφέρνουμε, αλλά ίσα ίσα που τα καταφέρνουμε. Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να αναζητήσουμε καλύτερες τεχνολογίες, χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Η πρόκληση είναι τεράστια. Ωστόσο, πρέπει να δούμε και πότε συμβαίνει η πρόκληση. Αν δείτε τα μοντέλα μας, θα δείτε ότι η μεγαλύτερη δυσκολία θα είναι στα επόμενα 10 χρόνια. Και όταν η SEC μας λέει ότι έχουμε ακόμα 10 χρόνια για να ε, λύσουμε το πρόβλημα, μας λέει ότι έχουμε 10 χρόνια για να βάλουμε μπροστά τις πολιτικές εκείνες οι οποίες θα, χρειαστεί, οι οποίες θα χρειαστούν μάλλον για να φτάσουμε στο 2050. Πρέπει δηλαδή να αναζητήσουμε την αναγκαία χρηματοδότηση, αναγκαίες επενδύσεις για να χρηματοδοτήσουμε την μετάβαση αυτή. Μετά θα πάνε πιο απλά τα πράγματα. Για τα επόμενα 10 χρόνια όμως αυτά τα 10 χρόνια είναι κρίσιμα. Τα επόμενα 10 χρόνια έχουμε για τα 10 χρόνια την, τις ρυθμίσεις, τις νομοθετικές ρυθμίσεις. Δεν, πρόκειται, βρίσκεται εκεί η πρόκληση, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να ασχολούμαστε και με το τι ακολουθεί. Πού θα ρίξουμε χρήματα στην έρευνα, τι είδου υποδομές θέλουμε να δημιουργήσουμε τι είδου πολιτικές, κρατικές ενισχύσεις, ανταγωνισμός, βιομηχανική πολιτική. Να τα κοιτάξουμε αυτά και να δούμε τι πρέπει, ποια πράγματα πρέπει να εμπλακούν στις πολιτικές αυτές. Να σταματήσω εδώ, πολύ σύντομα να πω το εξή CCS. Ναι, εμείς θεωρήσαμε ότι θα λειτουργήσει καλύτερα. Δεν πήγε καλά. Για τις ανανεώσιμες και εκεί τα πήγαμε, μάλλον και εκεί κάναμε λάθος υπολογισμό. Ευτυχώς όμως, γιατί πήγα πολύ καλύτερα από ό,τι είχαμε υπολογίσει. Αυτά τα μοντέλα αποδίδουν την πραγματικότητα όπως είναι σήμερα. Δεν είναι κανένα ιερό Ευαγγέλιο, δεν είναι καμία απόλυτη πρόβλεψη. Είναι μια σοβαρή ωστόσο προσπάθεια να δούμε πώς μπορεί να φαίνεται ο κόσμος, ποια μπορεί να είναι η εικόνα του κόσμου. Δεν ισχυριζόμαστε και καλά ότι έτσι θα είναι πράγματι ο κόσμος μίλησα για τη χρηματοδότηση, ένα μόνο, ε, μία μόνο κουβέντα για τα πυρηνικά. Αυτό το energy mix, το μείγμα ενέργεια είναι υπόθεση των χωρών μελών. Η πυρηνική ενέργεια υπάρχει. Δεν υπάρχει μια ένδειξη ότι οι περισσότερε χώρε μέλη θα εγκαταλείψουν πυρηνική ενέργεια. Και έτσι το παίρνουμε εμεί αυτό ω γεγονό, ότι υπάρχει δηλαδή. Και θα δούμε τι θα γίνει με το, με το μείγμα ενέργεια. Μάλιστα, σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλου και όλου. Εδώ λύγει το πρώτο πάνελ. Θα προσκαλέσω τώρα τους νέους τρεις πανελίστ, αφού ευχαριστήσω πρώτα όλους εσάς. Εσείς θα πρέπει να παραμείνετε κύριε Διευθυντά της Επιτροπής. Ας έρθει και η νέα προεδρεύουσα του επόμενου πάνελ. Να συνεχίσουμε λοιπόν ξεκινώντας το δεύτερο πάνελ και θα δώσω το λόγο αμέσως στον κύριο Ζερό Μέσεν από το Κλίμακτ. So, um, I'm coming Εκπροσωπώ την Climact και θα ήθελα να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα μιας μελέτης που κάναμε την προηγούμενη χρονιά. Πολύ γρήγορα θα ε, περάσω το περιβάλλον και τα γενικότερα ε, στοιχεία. Ε, δηλαδή, ναι, είναι δυνατόν μέχρι το 2050 να μειώσουμε τις εκπομπές κι άλλωστε το λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη στρατηγική της, αλλά θα πρέπει να ε, διευρύνουμε λίγο ε, αυτήν την βεντάλια των στοιχείων. Δεύτερον, εμείς μιλήσαμε, βασιστήκαμε σε κάποια σενάρια για την μελέτη μας ε, και επομένως λέμε ότι αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε μια καλή μετάβαση προς μηδενικές εκπομπές, τότε θα πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω μέχρι το 2000, να βάλουμε πιο φιλόδοξους στόχους. Επίσης, επίση υπάρχουν, ε, ε, το σενάριο αυτό είναι πιο ε, καλό και πιο αποτελεσματικό από ότι το business as usual σενάριο. το Ίδρυμα για το ε, Κλίμα ε, είχε ε, εκπονήσει έναν οδικό χάρτη, ένα χάρτη πορείας για το πώς θα πρέπει να είναι οι εκπομπές μέχρι το 2050. Βεβαίως υπάρχουν νέα στοιχεία, έχει πέσει πολύ το, στόχος, το κόστος συγγνώμη, των ανανεωσίμων, το IPCC ε, ε, λέει ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε κάτω από τους ε, δύο βαθμούς. Έχουμε εδώ σας δείχνω κάποιες μελέτες τις οποίες γνωρίζετε. Πολλές οργανώσεις και εμπειρογνώμονες έχουν συμβάλει μη κυβερνητικές οργανώσεις, εταιρείε, εμπειρογνώμονες κλπ. Και έχουμε αναπτύξει ένα μοντέλο το οποίο είναι ανοιχτό, διαφανές και διαθέσιμο επιγραμμικά έτσι ώστε αν θέλετε μπορείτε να ακολουθήσετε αυτό το μονοπάτι των μηδενικών εκπομπών. Το μοντέλο ακριβώς προσπαθεί να δει το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας, δηλαδή από τον τρόπο ζωής, lifestyle, τον τρόπο κατανάλωσης, ε, την κινητικότητα, την κατανάλωση καυσίμων, ε, τα κτίρια κτλ. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι χάρη στη μελέτη είχαμε τη δυνατότητα να δούμε πώς μπορούμε και με διάφορους τρόπους να επιτύχουμε τους στόχους μέχρι το 2050. Διάφοροι από, τους, ε, από τα πεδία, από τους τομείς ε, λοιπόν μας απασχόλησαν και θελήσαμε να δούμε ε, ε με ποιο τρόπο Mind that the demand side levers have been split into ε, νομίζω ότι θα πρέπει να μοιράσουμε, ε, να τα δούμε σε δύο κατηγορίες. Πρώτα απ' όλα ε, τα κοινωνικά στοιχεία, τα οποία έχουν τη γεννητικότητα κτλ και μετά ε, ε, ε, θα βάλουμε τους άλλους μοχλούς πίεσης που αφορούν ας πούμε τις υποδομές. Αν θέλετε να αλλάξει ας πούμε ο τρόπος της κινητικότητας για, προς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μα γι' αυτό χρειάζονται υποδομές. Επίσης λαμβάνουμε υπόψη κάποιες, κάποια στοιχεία που αφορούν την οργάνωση της κοινωνίας, κάποια άλλα στοιχεία, τεχνολογίες που αφορούν τις διαδικαστικές Εμμύχια. Ε, ε, ε, κλπ. Ανάλογα με, το στο, με τον τρόπο με τον οποίο διαβάζει κανείς αυτούς τους ε, μοχληρούς ε, μπορεί να ακολουθήσει τρία διαφορετικά σενάρια. Εδώ σας δείχνω τα, δια τα τρία σενάρια. Υπάρχει το σενάριο της τεχνολογίας όπου, όπου λαμβάνονται υπόψη και προωθούνται κυρίως όλοι οι μοχλοί που αφορούν ακριβώς αυτά τα στοιχεία και οι τεχνολογικοί μοχλοί μπορούν να μας φτάσουν μέχρι το μέσον της διαδρομής για τις μηδενικές εκπομπές. Υπάρχει το σενάριο της ζήτησης που μπορεί να αφορά ε, τον χώρο που έχει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ας πούμε για τις η οικονομία ε, για τα σπίτια κλπ. Και μετά υπάρχει το μοιρασμένο σενάριο. Ε, στα σενάρια αυτά οι περισσότεροι τομεί θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν και κυρίως ε, θα πρέπει να αφαιρεθεί ο, ο, ο άνθρακας μέχρι τα μέσα του αιώνα, μέχρι το 2050 δηλαδή, και από τη βιομηχανία και από τα κτίρια και από τις μετακινήσεις. Ε, μιλώντας πάντα ε, και έχοντας πάντα σαν κεντρικό στοιχείο του, τους ε, στόχους αυτούς ε, βλέπουμε ότι 25% μείωση μπορεί να γίνει ήδη με στοιχεία τα οποία τεχνολογικά και εμπορικά είναι ήδη διαθέσιμα. Και επιπλέον ε, έχουμε, ε, συγγνώμη, αυτό είναι 75% και το 25% που απομένει αφορά την τεχνολογική καινοτομία, αλλά όχι μόνο. Ε, μπορεί να υπάρξει καινοτομία όσον αφορά τα business models, τα επιχειρηματικά μοντέλα, όσον αφορά την κυκλική οικονομία, όσον αφορά, ας πούμε, την λειτουργική οικονομία, όπου όλα τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν στον μεγαλύτερο δυνατό κύκλο ζωής. Αυτό προϋποθέτει όμως έναν νέο τρόπο ε, πώλησης και διαμοιράσματος των στοιχείων. Επομένως, μελετώντας τα σενάρια αυτά, μπορούμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο ε, μπορούμε να προχωρήσουμε μέχρι το 2050. Στην μπλε γραμμή βλέπουμε ε, την μείωση που μπορεί να επιτευχθεί μέσω των τριών ε, οδών που ανέφερα προηγουμένως. Μπορείτε όμως να διαπιστώσετε ότι η πρόθεση της Κομισιόν για μείωση 45% μέχρι το 2030 εξακολουθεί να είναι υψηλότερος ο στόχος από τα σενάρια τα οποία εμείς μοντελοποιήσαμε. Και βεβαίως όσο περιμένουμε ε, τόσο πιο δύσκολα θα γίνει η μετάβαση. Τούτων ελεγχθέντων μέχρι το 2030, όποια οδό και αν έχει επιλέξει κανείς, ε, θα ε, πρέπει να έχουν γίνει οπωσδήποτε, να έχουν ληφθεί οπωσδήποτε κάποιες ε, αποφάσεις. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει σταθεροποιηθεί η ζήτηση των μεταφο... στον τομέα των μεταφορών. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε καινοτομία στις οικοδομές. Θα πρέπει να έχουμε φτάσει τουλάχιστον στο 50% της ενέργειας από ανανεώσιμε ε, πηγές ενέργειας, ηλιακή κλπ. Θα πρέπει επίσης να έχει αλλάξει ε, η πολιτική χρήση γη και θα πρέπει να έχει προσαρμοστεί στο κλίμα. Θα πρέπει να δούμε επίσης ε, και το κόστος όσον αφορά τις επενδύσεις. Ε, όταν πρέπει να ε, πληρώσει κανείς για νέο σχεδιασμό θα πρέπει να προσθέσουμε σε αυτό το κόστος των καυσίμων και τέλος την λειτουργία και την συντήρηση. Επομένως θα πρέπει να γίνει μια, ένας καλός υπολογισμός του κόστους ωφέλους. Εδώ βλέπετε στα αριστερά το σενάριο ΡΕΦ. Ε, το οποίο ε, αναφέρει, αναφέρεται σε κάποια κόστη τα οποία ανεβαίνουν λίγο αλλά ε, όχι πάρα πολύ κυρίως όσον αφορά σαν σε κυρίως όσον αφορά την αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας, ενώ το σενάριο net zero δεξιά βλέπετε ότι υπάρχει μια σταθερή, ένα σταθερό ποσοστό. Ε, επίσης έχουμε ένα άλλο ε, σενάριο ε, σχέσεις ανάμεσα στην τεχνολογία και την ενέργεια που μπορεί να δώσει χαμηλότερα ε, μπορεί να δώσει ε, υψηλότερες αποδόσεις ενώ στο σενάριο της τεχνολογίας φτάνοντας περίπου στο 2030 ε, μπορεί να έχουμε καλά αποτελέσματα αλλά η ενεργειακή η αποδοτικότητα δεν θα είναι τόσο καλή. Όταν αν δει κανείς το, την μέση δαπάνη αναέτος που θα πρέπει να έχουμε για κάθε σενάριο παραπάνω από δύο δις ε, στο πρώτο σενάριο, λιγότερη μέση ετήσια δαπάνη για το shared ε, σενάριο και οπωσδήποτε υψηλότερη για το τρίτο σενάριο. Ε, όμως η διαφορά, λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω, είναι σαφώς μικρότερη από ότι η ζημιά που μπορούμε να περιμένουμε, να αναμένουμε όσον αφορά το, την κλιματική αλλαγή και δεξιά ε, βλέπετε ακριβώς την ε, αυξανόμενη επένδυση που θα πρέπει να γίνει καθώς επίσης και την επιστροφή ε, και τη σχέση κόστους οφέλους όσον αφορά ε, την αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση κτλ. Ε, ε, όταν λέμε net zero, καθαρά μηδενικό σενάριο, σημαίνει ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να βρούμε έναν νέο τρόπο, ε, πιο πολύ διαφορετικό από ό,τι στα προηγούμενα σενάρια για την παραγωγή ενέργειας και σε όλα τα σενάρια για το 2030 το κόστος αυτό είναι χαμηλότερο από ότι το κόστος αναφοράς. Muchas gracias. A continuación mm, tiene la palabra Mrs. Η κυρία Ward ε, θα έχει τώρα τον ε, λόγο, η οποία ε, είναι επικεφαλής στρατηγικής στην IIGCC. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας απευθύνω το λόγο. Όσοι λοιπόν είναι εξοικειωμένοι με τις, τους επενδυτές για την κλιματική αλλαγή, 130 είμαστε περίπου. Και μερικά είναι και τα μεγαλύτερα ε, επενδυτικά συνταξιωτικά ταμεία από 11 χώρες, 22 δις. Ε, τρεις είναι η επένδυση. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να κινητοποιούμε κεφάλαιο για ένα ε, βίωνο μέλλον. Σήμερα θα μιλήσω για την υποστήριξη της δήλωσης της ε, Κομισιόν και για το σχέδιο ψηφίσματος του Κοινοβουλίου. Ακούσαμε πάρα πολλά σήμερα για τις επενδύσεις. Εγώ θα ήθελα να κάνω λίγο πίσω και να δούμε γιατί είναι σημαντική η κλιματική αλλαγή για τους επενδυτές. Ε, τι είναι εκείνο που είναι μια πολιτική που αξίζει να γίνονται επενδύσεις Πρώτα απ' όλα λοιπόν, οι επενδυτές ενδιαφέρονται για την κλιματική αλλαγή γιατί πολλοί επενδύουν σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε όλους τους τομείς, σε όλες τις χώρες. Άρα δηλαδή ε, εκτίθεται κανείς και σε συστημικές αλλαγές όπως είναι, η κλιματική αλλαγή. Μοιάζει να ελέγχεται η κατάσταση, να ε, μπορούν να προβλεφθούν αποτυχημένα κεφάλαια. Υπάρχουν όμως και επενδυτικές ευκαιρίες, κυρίως όσον αφορά τη μετάβαση σε ε, οικονομία χωρίς ε, άντρακα, Άρα δηλαδή για αυτούς τους λόγους πάρα πολλοί επενδυτές ε, είναι ιδιαίτερα ενεργοί στην κλιματική αλλαγή. Παραδείγματο χάνει ενεργειακέ επενδύσει από 37% σε 43% από το 2014 μέχρι το 2016 επενδύσει σε τομεί χωρί άντρακα. Η έρευνα που έγινε ε, το 2017 έδειξε ότι το 97% όσων απάντησαν στην Ευρώπη σκέπτονται να αυξήσουν τις επενδύσεις λόγω κλιματικής αλλαγής. Επίσης, οι επενδυτές δεσμεύονται να αναφέρουν τους κινδύνους ε, μέσα από τις, ε, την αποκάλυψη των οικονομικών και τέλος έχουμε μία παγκόσμια πρωτοβουλία όπου όπως σας είπα δολάρια τώρα επενδύονται από από τις επενδυτικές εταιρείες. Όμως όλα αυτά θα μπορούσαν να καθυστερήσουν με βάση τα οικονομικά πλαίσια που υπάρχουν. Γιατί ε, τα προγράμματα ε, θέλουν να γνωρίζουν κατά πόσον οι επενδυτές μπορούν να αξιολογήσουν τους κινδύνους και να επενδύουν σε δυνατότητες, σε οικονομίες χωρίς άνθρακα. Το 2017 κάναμε μία μελέτη. Περίπου το 80% των μελών είπαν ότι υπάρχει κάποια ανασφάλεια. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους επενδυτές. Και είπαν τα μέλη μας ότι θέλουν σαφήνεια για το πώς οι κυβερνήσεις και οι ενωσιακοί ε, θεσμοί ε, σκοπεύουν που να εφαρμόσουν τη Συμφωνία του Παρισιού. Άρα δηλαδή ποια είναι η καλή πολιτική για τους επενδυτές. Οι χώρες που είναι υπέρ του χαμηλού άνθρακα και που εφαρμόζουν μακροχρόνια προγράμματα είναι οι χώρες εκείνες που κατόρθωσαν να κάνουν επενδύσεις. Ε, η ανταπόδοση, διαφανής, ε, διαφανής πολιτική, αυτά προσελκύουν το κεφάλαιο. Βλέπετε εδώ ε, τις τέσσερις πολιτικές προϋποθέσεις που ισχύουν για μας σε γενικέ γραμμέ, οι επενδυτέ αναζητούν πρώτα ένα πολιτικό περιβάλλον το οποίο δεσμεύεται σε μείωση του άνθρακα και αυτή η δέσμευση βασίζεται σε μια πολύ καλή συνεννόηση για του περιβαλλοντικού κινδύνου και τι ευκαιρίε. Δεύτερον, πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για να καλύπτονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι. Μετά, να υπάρχει ένα σταθερό νομοθετικό πλαίσιο, μειών του κινδύνου για του επενδυτέ, ε, υπάρχουν προβλέψιμα κέρδη, ε, τεχνολογία χαμηλού άνθρακα στην αγορά στο πλαίσιο προγράμματος και απόρριψη των ε, αναδρομικών ε, και οπισθοδρομικών αλλαγών. Αυτά να εντάσσονται σε μια πολιτική που να είναι συνεπής με την ε, συνδυάσκεψη του Παλισιού. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Σε γενικές γραμμές η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε σταθερά θεμέλια. Οι επενδυτές χαιρέτησαν την δήλωση της Κομισιόν πέρυσι και αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 30, εκεί αναφέρεται ότι 130 δισεκατομμύρια δολάρια χρειάζονται κάθε χρόνο μέχρι το 2030 ε, για τις ανανεώσιμε πηγές και για να νοωθεί και να νοηθούν υποδομές. Τεράστια ευκαιρία, αλλά για να προσελκυθεί τόσο μεγάλο κεφάλαιο, οι πολιτικοί θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι η πολιτική θα ασχολείται με τα εξή. Πρώτον, θα επιβεβαιώνει μακροχρόνιο στόχο απομάκρυνση του άνθρακα, να φτάσουμε σε μηδενικές εκπομπές, το αργότερο μέχρι το 2050. Επίσης, να αναγνωριστεί ότι ορισμένα κράτη-μέλη μπορεί να θέλουν αυτό να το πετύχουν νωρίτερα, ανάλογα με τις συνθήκες. Και ε, ως εκ τούτου πρέπει να είναι δυνατόν να αναθεωρηθεί όλο αυτό σε μελλοντικέ επιστημονικές μελέτες. Δεύτερον, όλη αυτή η προσέγγιση πρέπει να είναι ολιστική όλοι οι παράγοντες να παίζουν ρόλο, προγράμματα δηλαδή για το πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να περιορίσει τις εκπομπές σε όλου του τομείς, περίπου στο 0, το αργότερο μέχρι το 50. Παραδείγματο χάρη, ε, φτάνοντας σε ένα σύστημα ε, το οποίο θα στηρίζεται και αποκαλεί τιμή του άνθρακα. Να υπάρχει στρατηγική ε, που να απορροφά τον άνθρακα που, δεν έχει, που, εκπέμπεται ακόμα. Πιστεύουμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε τους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να είναι ε, σε αρμονία με τους στόχους του 50 και τη Συμφωνία του Παρισιού. Επίσης, ε, το νομοθετικό πλαίσιο να επιτρέπει έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία και να εντοπίζει που χρειάζονται περισσότερα κεφάλαια για να στηριχθεί η ανάπτυξη. Για το μέλλον πρέπει να αναφέρεται πώς οι αποφάσεις θα αξιολογηθούν έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης εναρμόνιση με τη στρατηγική για το 2050. Και τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα στηρίζει τον προσανατολισμό προς τον οποίο κατευθύνονται όλοι αυτοί οι στόχοι, έτσι ώστε να υπάρχει μια καλή μετάβαση ε, προς μια οικονομία χαμηλού άνθρακα. Τρίτον, η στρατηγική πρέπει να συνεχίσει ε, να υπολογίζει τους κινδύνους. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούν να υπάρξουν σημαντικά σημαντικές ζημιές για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρέπει να ξεχνάμε να επενθυμίζουμε τι ακριβώς αντιμετωπίζουμε. Ε, η IGCC καλωσορίζει το σχέδιο του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί εκεί αναφέρεται ότι πρέπει να υπάρχει προβλεψιμότητα, συμπληρωματικότητα και ε, περιεκτικότητα. Και εμεί ε, καλωσορίζουμε την ευκαιρία να έχουμε περαιτέρω συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να μπορούμε να μοχλεύσουμε τι επενδύσει του ιδιωτικού τομέα. Ε, αυτό ισχύει και για του ιδιώτε και για τα κράτη-μέλη. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι να επαναλάβω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελε σε παγκόσμιο επίπεδο να είναι η πρώτη δύναμη που θα δείξει πώ μπορεί κανεί να επιτύχει του ε, στόχου του Παρισιού με μηδενικέ εκπομπές. Ε, υπάρχουν επενδυτικά δίχτυα και επενδυτικές ευκαιρίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού και όλοι αυτοί μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο μαζί και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πραγματικά τα μάτια του κόσμου είναι στραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δει πώς θα προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις και όλα βασίζονται στην επιτυχία της στρατηγικής του 2050. Για να ολοκληρώσω, υπάρχει ένα όραμα Υπάρχουν βέβαια κίνδυνοι που έχουν μειωθεί ή επενδυτικές ευκαιρίες έχουν προκύψει από αυτή την ανάγκη του να υπάρχει χαμηλή χρήση άνθρακα υπάρχουν και πολλά κοινωνικά, περιβαλλοντικά και άλλα ωφέλη. Άρα δηλαδή τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να καταδείξει στους εταίρους ότι μια πράσινη οικονομία μέχρι το 2050 είναι εφικτή και εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και με όλους τους άλλους εταίρους μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί δεν ξεπεράσατε και το χρόνο σας. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Κλέρ Ρουμέ από την Energy Cities και την ε, Σύμβαση των ε, Δημάρχων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το καλό ε, που έχει κάποιος που μιλάει τελευταίος είναι ότι δεν χρειάζεται ε, να επαναλάβει πράγματα τα οποία έχουν ήδη ακουστεί και επομένως ε, μπορεί να περιοριστεί σε αυτά που ακούγονται πρώτη φορά. Στο πάνελ εδώ έχει αναφερθεί το δυναμικό των ε, πόλεων. Εγώ θα ήθελα να πω ότι έχουν ήδη κάνει οι πόλεις και τι σκοπεύουν να κάνουν που, ε, πράγματα δηλαδή που ευθυγραμμίζονται με αυτά που ε, λέει η, η Κομισιόν και αυτά που προτείνει μέσω της μακροχρόνιας ε, ε, στρατηγικής. Ε, μπορούμε να επιτύχουμε λοιπόν τις μηδενικές εκπομπές και ας προχωρήσουμε να καταφέρουμε να το κάνουμε. Βεβαίως, όπως είπε και η Κομισιόν προηγουμένως, αυτό δεν μπορούν να το κάνουν οι Βρυξέλλες ε, μόνες τους. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι τομείς, όλοι οι πρωταγωνιστές σε κάθε διαφορετικό επίπεδο διακυβέρνησης ευθυγραμμίζονται όλοι για να διασφαλίσουν αυτό το αποτέλεσμα. Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ ε, δεν αναγνωρίζουμε αρκετά το γεγονός ότι τα 4-5 τελευταία χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν αλλάξει το τοπίο της ενέργειας και αυτό είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό γιατί και εμείς ε, σαν ε, τοπικοί παράγοντες δεν μπορούσαμε να πάρουμε κάποιες δράσεις γιατί μέχρι τότε δεν μας αναγνώριζαν αυτό το καθεστώς του πλήρους ε, ε, πρωταγωνιστή ας πούμε. Ε, και αυτή τη στιγμή μιλάμε για αποκεντρωμένη διακυβέρνηση και παραγωγή ενέργειας. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα και το θέμα της διακυβέρνησης επίσης μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μπορούν να σχεδιαστούν πολιτικές από κάτω προς τα πάνω και ε, να, χρησιμοποιήσει, ε, να χρησιμοποιηθεί όλο το δυναμικό ε, των τοπικών δυνατοτήτων. Για να είμαι σύντομη το πιο σημαντικό σημείο ή στοιχείο είναι ο, για το κλίμα στις Βρυξέλλες και αλλού, ε, αυτές δηλαδή που οργανώνονται σε όλες τις χώρες. Ε, ε, την προηγούμενη Κυριακή είχαμε μια μεγάλη πορεία για το κλίμα των μαθητών και το Δημοτικό Συμβούλιο των Βρυξελών εξέδωσε ειδικό ψήφισμα βάσει μιας κατεπίγουσας συζήτησης όπου αναφέρεται ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να επιταχυνθεί η υλοποίηση του δικού τους ε, ε, σχεδίου δράσης για την ενέργεια. Δηλαδή αφουγκράζονται τα όσα συμβαίνουν ε, στο δρόμο και θέλουν να προωθήσουν σε τοπικό επίπεδο επιταχυμένες διαδικασίες. Αυτό αυτό δεν αντιτίθεται ε, μάλλον ήθελα να πω ότι κινήματα όπως ας πούμε τα κίτρινα γυλαίκα δεν αντιτίθενται ε, σε αυτή την επιταχυμένη διαδικασία. Ε, είχαμε στην Γαλλία με τα κίτρινα γυλαίκα μια διάσκεψη για την ενεργειακή μετάβαση και προέκυψε σαφώς ότι αυτό που θέλουν είναι ε, η ε, διαμοιρασμένη ας πούμε μετάβαση, share transition, ε, δηλαδή εάν όλοι κατανοούν με τον ίδιο τρόπο την κατάσταση, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε στην ενεργειακή μετάβαση. Δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε ας πούμε στην μετάβαση εάν φόρος, θα, φόρος μετακίνησης αφορά μονάχα τις χερσαίες μεταφορές ας πούμε και όχι τις αεροπορικές ή τις θαλάσσιες. Οι πολίτες μας τα βλέπουν αυτά ε, και ε, πλέον ε, απευθύνονται, στρέφονται στους τοπικούς ερετούς άρχοντες στους, έτσι ώστε να συζητήσουν για τα θέματα αυτά και να εκδηλώσουν την ανάγκη για ανάληψη δράσης. Στην Φιλανδία, ας πούμε, έχει στόχο ε, για μηδενικές εκπομπές, οικονομία μηδενικών εκπομπών μέχρι το 2013. Ναι, και η πόλη του Ελσίνκη προσπαθεί ε, να εφαρμόσει στην ε, ε, τοπική οικονομία αυτόν τον στόχο, τον εθνικό στόχο για το 2035. Περί αυτού πρόκειται λοιπόν η μακροχρόνια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει το πλεονέκτημα να θέτει ένα γενικό πλαίσιο, αλλά εμείς εάν θέλουμε πραγματικά να επιτύχουμε αυτό το φιλόδοξο σχέδιο των μηδενικών τότε ο κάθε εμπλεκόμενος σε κάθε επίπεδο θα πρέπει να καλύψει τη δικιά του αποστολή εντός αυτού του κοινού και διαμοιρασμένου πλαισίου. Εδώ σας δίνω ένα παράδειγμα ε, του Παρισιού. Ξέρετε ότι μέχρι το 2050 μπορεί να ελευθερωθεί από τον άνθρακα ε, το Παρίσι. Σε κόκκινο βλέπετε την ε, διοίκηση του Παρισιού. Δηλαδή είναι ένα πάρα πολύ μικρό ε, κομμάτι των ε, εκπομπών στο Παρίσι. Μονάχα ένα μικρό ε, κλάσμα του 2% εξαρτάται από την από την κεντρική κυβέρνηση. Τα υπόλοιπα αφορούν την τοπική ε, αρχή που μπορεί να αλλάξει τον μεταβολισμό ε, της ε, πόλης. Και σας λέγω ότι ομόφωνα έγινε δεκτός ο οδικός χάρτης, αυτός ο χάρτης πορείας του Παρισιού προς τον στόχο των μηδενικών εκπομπών. Και επομένως σε τοπικό επίπεδο μπορεί να αναλυθεί ε, Ίσως να κάνω και κάποια επιπλέον σχόλια, να σας πω ε, τι απαιτείται για τα επόμενα βήματα. Βεβαίως έχουμε την μακροχρόνια στρατηγική, η οποία, την οποία ενστερνίζονται όλες, ε, όλα τα θεσμικά όργανα, αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρξει μια ευθυγράμμιση όλων των φορέων ας πούμε, στο Μάντσεστερ έχουν δημιουργήσει την λεγόμενη Climate Change Board ε, που, ε, ε, θέλει να, που μελετά την ευθυγράμμιση όλων των τοπικών πολιτικών με τον στόχο αυτό για το κλίμα και για τις εκπομπές. και ε, ε, πιστεύουμε ότι και στα πλαίσια του επομένου προγράμματος Horizon 2020 στο σκέλος της έρευνας θα πρέπει οπωσδήποτε να μελετηθούν τα τοπικά μοντέλα τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στη συνολική αλλαγή. Αυτά ήθελα να πω, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Ε, να σας πω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας ότι η τεχνολογία υπάρχει ήδη δεν χρειάζονται ε, τρομερές ε, πρόοδοι όσον αφορά την τεχνολογία. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε έναν τρόπο να μειώσουμε στο 50% τις ενεργειακές μας ανάγκες, πράγμα που προϋποθέτει βεβαίως διαφορετική οικονομική αντιμετώπιση, άλλα οικονομικά μοντέλα ε, και οπωσδήποτε να πούμε ότι σε τοπικό επίπεδο οι δήμαρχοι είναι έτοιμοι να αναλάβουν δράση και δεσμεύσεις για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η πρόεδρος Αγιούσο. Να περάσουμε τώρα αμέσως στην ε, ώρα των ερωτήσεων. Υπάρχει κανείς που επιθυμεί να ερωτήσει. No, pues en κάσο, Ορίστε κύριε Βόλκεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σύντομη ερώτηση. Μόλις μιλήσαμε τώρα για το Fight for Future, για, για τις των μαθητών και μαθητριών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, που βρίσκω πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που ε, κάνουν οι νέοι άνθρωποι, ε, κατεβαίνουν στους δρόμους δηλαδή και βλέπω και με πόση σαφήνεια απαιτούν επιτέλους να αναλυθεί κάποια δράση. Δηλαδή εμείς οι πολιτικοί να διασφαλίσουμε ότι η υπαρξιακή τους βάση δεν θα καταστραφεί. Από τη δική σας σκοπιά υπάρχουν ιδέες ή προτάσεις για το πώς μπορούμε να προσετριστούμε τους νέους αυτούς ανθρώπους που επιθυμούν να κάνουν κάτι. Δεν θα ήταν σωστό να προβληματιστούμε σχετικά για το πώς μπορεί να διασφαλίσει κανείς, για παράδειγμα, ότι η αντιπροσώπευση ή η εκπροσώπηση των γενεών ε, υλοποιείται. Θεωρείτε ότι πρόκειται για μια καλή ιδέα. Ο κύριος Μπράνιν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε ερωτήσεις. Αποθήκευση οξυδίων του άνθρακος, που συζητήθηκε στο, στο προηγούμενο γύρο ερωτήσεων. Είχαμε πάει και προ δύο-τριών ετών στην Ορβηγία για να δούμε ε, μια δοκιμή κλίμακος. Και το ίδιο συμβαίνει και στον Καναδά, σε μεγάλη κλίμακα. Υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το κόστος, αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο μείγμα ενέργειας. Θα ήθελα να, πείτε, να κάνετε κάποιο σχόλιο για το CCS, αποθήκευση δηλαδή οφείων του ανθρακός. Τώρα, δεύτερο, για τη στέγη. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο το βασικό είναι να εξοπλιστούν εκ των υστέρων τα υφιστάμενα ακίνητα. Βέβαια, το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να μην είναι πια μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι μια χώρα όπου υπάρχει έλλειψη στέγης και η Βρετανική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα χτίζει 300.000 ακίνητα 300, σπίτια, κατοικίες τον χρόνο. Και σε άλλες χώρες όπως Ινδία, Μεξικό, Βραζιλία, εκεί επίση υπάρχει κρίση στέγης. Αν όλες αυτές οι κατοικίες φτιαχτούν με παραδοσιακό τρόπο από τούβλα, τσιμέντο και ατσάλι, τότε καταστρέφουμε οποιαδήποτε πιθανότητα να πετύχουμε τους στόχους, διότι ε, αποδίδουν όλα αυτά, όλες, η παραγωγή, η παραγωγή, η παραγωγή όλων αυτών των υλικών ή ούτως ή άλλως οξύδια του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και ξαναρχόμαστε στα ίδια. Θα χρειαστεί λοιπόν να δώσει ε, όθηση ε, σε άλλα υλικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ξυλία. Να χτίζονται δηλαδή ε, κατοικίες από ε, κατελεσμένη ξυλία. Πόση σημασία αποδίδεται στην πρόθεση αυτού του σχεδίου. Θα δώσω τώρα το λόγο. Α, στην κυρία Νταλή θα δώσω το λόγο. Σύντομη ερώτηση. Λέχθηκε ότι οι επενδυτές χρειάζονται μηνύματα και ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι μόνο πρόκληση ή κίνδυνο, αλλά υπάρχουν και οικονομικέ ευκαιρίε. Αυτό μπορεί να προσφέρει νέε επιχειρηματικέ ευκαιρίε και να δημιουργήσει νέου οικονομικού τομεί από οι τομείς τη οικονομίας. Από την εμπειρία σα. Πώ βλέπετε οι επιχειρήσει να αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή ω κίνδυνο και ω πρόκληση. Νομίζω ότι κάνουν αρκετά πράγματα και ε, τι προτάσει μπορείτε να κάνετε ή τουλάχιστον Ποιε προτάσει θα θέλατε να δείτε να καταδείχνετε σε ό,τι αφορά τα επιχειρηματικά σχέδια και επίσης το πώς η βιομηχανία αντιμετωπίζει την πρόκληση αυτή, ώστε να μην είναι μόνο πρόκληση αλλά και ευκαιρία. Εσείς κύριε Πετιτσιόνε τώρα για να μπορέσετε να απαντήσετε. Thank you, Madam uh, Λοιπόν, δεν έχω πολλά να προσθέσω, απλά να υπογραμμίσω ορισμένα σημεία και να αναφερθώ σε αυτό που ρώτησε η κυρία Ντάλη στο τέλος. Ε, πραγματικά εντυπωσιάστηκα από τις τέσσερις απαιτήσει ε, που έχουν θέσει οι επενδυτές, όπως ανέφερε και η κυρία Γουόρντ. Τρεις εξ αυτών ισχύουν για οποιαδήποτε μορφή επένδυση. Μόνο μία προϋπόθεση είναι καινούργια. Είναι η πολιτική δέσμευση για την χρήση ε, χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Ε, τον τελευταίο καιρό μιλώ συνέχεια με επενδυτές, βιομηχάνους ε, και το ακούω μέχρι κοπόσεως που λένε δώστε μας το πλαίσιο, πέστε μας ποιοι είναι οι στόχοι και μετά γίνεται λόγος ότι δώστε μας υποστήριξη, καθορίστε ένα πλαίσιο και μετά μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση. Αλλά το σημαντικότερο όλων είναι θέλουν να μάθουν κατά πόσον έχουμε πράγματι στόχο. Και ποιο είναι αυτό ο στόχο. Νομίζω αυτό λείπει. Στην Ευρώπη είμαστε αρκετά καλοί ε, στις ε, σταδιακές πολιτικές και αν δείτε λιγάκι την εξέλιξη της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια, ε, καλά τα καταφέραμε. Όμως κανονικά ε, το χρονοδιάγραμμα είναι πρόβλημα. Ε, έχουμε πρόβλημα με τις καθυστερήσεις. Εδώ έχουμε πραγματικά καταληκτική μερομηνία που είναι θέμα ζωής και θανάτου. Πρέπει να αποφασίσουμε ε, Ποιε είναι οι προποθέσει και μετά να προχωρήσουμε την τρίτη χρονιά, γιατί αλλιώ ε, χάνουμε το χρόνο μας. Νομίζω ότι για μένα, όπως σα είπα και προηγουμένω, ε, αυτό κατ' ουσίαν είναι επενδυτική πρόκληση. Δεν είναι θέμα κόστου, δεν πληρώνουμε για να λύσουμε τα προβλήματα του παρελθόντο. Πρέπει κάπως να βρούμε του πόρους. Πρέπει να με τους απαραίτητους πόρους και οι άνθρωποι και εκείνοι για να επενδύσουν θέλουν να ξέρουν τι θέλουμε να κάνουμε. Αυτό για μένα είναι καθοριστική σημασία. Είδαμε το σχέδιο ψηφίσματος του Κοινοβουλίου. Ε, με μεγάλη μας χαρά διαβάσαμε αυτά που περιλαμβάνει, παρά τη διάσταση απόψεων για μεμονωμένα θέματα, για τους στόχους, φιλοδοξίες. Χαίρομαι που υπάρχει συνένεση ε, στο Κοινοβούλιο. Για τη τελική ανάλυση πιστεύω ότι αυτά θα γίνουν όλα αυτόματα. Εμείς θέλουμε να υπάρξει συζήτηση. Θέλουμε να γίνει μια όσο πιο σκληρή συζήτηση γίνεται, γιατί σε τελική ανάλυση χρειαζόμαστε ένα στόχο, τον οποίο θα τον υποστηρίζουν όλοι ανεπιφύλακτα. Μόνο έτσι θα έχουμε την πολιτική υποστήριξη για να προχωρήσουμε. Γιατί τα επόμενα δέκα χρόνια ε, θα απασχοληθούμε πάρα πολύ με το να εντοπίζουμε τις δράσεις που προέκυψαν από αυτούς τους στόχους. Πολύ ωραία. Κύριε Πετιτσόνε, τώρα το λόγο έχουν οι τρεις μας ομιλητές για να απαντήσουν σε αυτές τις ερωτήσεις. Και θα ακολουθήσω την ίδια σειρά όπως και προηγουμένως. Να απαντήσω για τις τεχνικές ερωτήσεις. Ο γιος μου την προηγούμενη Πέμπτη την κοπάνισε από το σχολείο για να πάει να διαδηλώσει στις Βρυξέλλες. Δεν λέω τίποτα προσωπικά γι' αυτό, αλλά α μην αργήσουμε και α αρχίσουμε να κάνουμε κάτι. Είναι διαθέσιμε οι τεχνολογίε, όπω είδατε και στην παρουσίαση. Δεν υπάρχουν πολλέ επιλογέ no regret. Στα διάφορα σενάρια έχουμε μοντέλα και ε, αυτά μας υπαγορεύουν πολλού λόγους για να μην περιμένουμε άλλο. Τώρα, για το CCS, ε, αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακο. Ίσως είναι σωστό να επισημάνουμε ότι εμείς δεν προτείνουμε μία τεχνολογία, ούτε προτιμώ μία τεχνολογία, ούτε δίνουμε αναλύσεις κόστους ωφέλους σε ένα ε, βέλτιστο σενάριο. Έχετε τη δυνατότητα με τα μοντέλα να κάνετε ε, προσωμιώσεις ε, σενάριων με το CCS και χωρίς. Είναι δυνατόν να γίνουν προσωμιώσεις σενάριων σε net zero χωρίς CCS, αλλά αυτό βέβαια σημαίνει ότι θα κάνουν μεγαλύτερη ε, προσπάθεια η άλλοι τομείς και ιδίως οι τομείς της ζήτησης. Ε, μιλήσατε εσείς για το παράδειγμα των κτηρίων. Για το ερώτημά σας σχετικά με την κατασκευή στέγης, αυτό είναι ζήτημα πολιτικής περισσότερο και ξεφεύγει κάπως από το πλαίσιο των όσων παρουσιάζουμε σήμερα. Προτιμώ να μην απαντήσω. Η υποκατάσταση υλικών τώρα, με υλικά, μάλλον η αντικατάσταση υλικών κατασκευής με ναι, άλλα, όπως για παράδειγμα η ξυλία αντί του χάλιβα και του τσιμέντου. Ασφαλώς και αποτελεί ε, ένα είδος μοχλού που μπορεί να συζητηθεί και να αναλυθεί περισσότερο στο μέλλον. Και αυτό περιλαμβάνεται στα σενάρια. Ξαναλέω όμως ότι είδαμε επίσης ότι πρόκειται για πρόκληση για τους επενδυτές, όπως είπε και ο ίδιος ο κύριος Πέτριτσόνε. Είδατε πως υπάρχουν φάσεις επενδύσεων και φάσεις αναμονής των ε, ωφελιών. Ευχαριστώ. Απαντώ πρώτα στην κυρία Ντάλη για τις επενδύσεις. για την προσέγγιση των εταιριών στην κλιματική αλλαγή. Όπως είπα πριν, πρόκειται για μια νέα δράση 100 συν που ζητεί από τους επενδυτές να δραστηριοποιηθούν περισσότερο. Βλέπουμε επιτυχία σημαντική από την πρωτοβουλία αυτή. Ως παράδειγμα, πρόσφατες, πρόσφατες από τη Shell και ExxonMobil μετά από πίεση των επενδυτών επί των εταιριών αυτών. Ακόμα δεν έχουν γίνει περισσότερα πράγματα, γι' αυτό και η πρωτοβουλία αυτή προβλέπει μια πενταετή διάρκεια, όπου οι επενδυτές συζητούν ειλικρινά, παρασκηνιακά, με διοικητικά συμβούλια, με τους καταπιστευματούχους για να δουν στο τέλος της πενταετίας αν έγιναν αρκετά πράγματα ώστε να ληφθούν κάποιες δύσκολες άλλωστε αποφάσεις για το μέλλον των επιχειρήσεων αυτών. Υπάρχει ταυτόχρονα βέβαια και πίεση από το κοινό με ψηφίσματα κλπ. Και εκεί χρειάζεται να συντονιστούν και αυτά. Σε ό,τι αφορά το τι χρειάζεται περισσότερο να γίνει τώρα, εμείς συστήνουμε ορισμένα πράγματα στις επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα να διασφαλίσουν ότι θα είναι ενήμερο το Διοικητικό Συμβούλιο και οι καταπιστευματοδόχοι τραστείς δηλαδή σχετικά με τις ανάγκες του κλίματος για να τις περιλάβουν στις ε, διαδικασίες ε, λήψεως αποφάσεων, να μην παραμένουν δηλαδή κάπου σε ένα σιλό ξεχωριστό οι γνώσεις και οι αποφάσεις αυτές. Χρειάζεται δηλαδή να εξετάσουν τους ρόλους που παίζει η ηγετική ομάδα και πώς αυτή η διακυβέρνηση μετά καταλήγει να φτάσει σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης της ε, επιχειρήσεως. Επίσης, διέται ε, ε, ε, κοινά γνωστή αυτή η πληροφόρηση, ώστε να φτάσει και ως τους μετόχους. Αυτά είναι ορισμένα από τα πράγματα που προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε με τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Για να απαντήσω σύντομα σε άλλες ερωτήσεις τώρα, είχε ενδιαφέρον ότι αναφέρθηκε η κατασκευή στέγης στους δικούς, για τους δικούς επενδυτές στέγη και ε, ακίνητα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Και οι επενδυτές μας κάνουν προσπάθειες και στην ανακαίνιση και στις ε, νέες κατασκευές κατοικιών με ε, θεσμούς όπως ΙΦΕ, με δάνεια για, που χορηγούνται σε ανθρώπους οι οποίοι επιθυμούν να χτίσουν με καινοτόμες τεχνικές και ούτω καθεξής. Και αυτά και μέσα στα πλαίσια τη διαπραγμάτευση για την σχετική οδηγία. Και συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε και με τι χώρε μέλη για το σύστημα αποθήκευση οξυδίων του άνθρακο. Από τότε που εκδόθηκε η έκθεση τη IPCC, έχω δει ότι οι επενδυτέ ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για την διερεύνηση ε, των σχετικών δυνατοτήτων. Είδατε και αυτό που είπατε εσείς, οι δοκιμέ κλίμακο και επενδύουν περισσότερο σε αυτές τις τεχνολογίες, αλλά υπάρχει ακόμα δρόμος που πρέπει να καλυφθεί. Σε ό,τι αφορά τις νέες και τους νέους και τις ε, αξιώσεις τους, οι δικοί μας ε, βέβαια επενδυτές είναι στα αξιωτικά ταμεία, τα έχουν περιλάβει αυτά στα business model. Αλλά αυτό που ενδιαφέρονται είναι βέβαια να μεγιστοποιήσουν το όφελος για τους ε, μετόχους τους, δηλαδή τους συνταξιούχους. Αυτά θα απασχολήσουν τους νέους στο μέλλον. Εάν επιτευχθεί η στρατηγική 2050, αν επιτύχει δηλαδή, θα αντιμετωπίσει και κάποιε από τις απαιτήσει των νεότερων γενεών. Uh, θα είμαι πολύ σύντομη. Όσον αφορά τις οικοδομές υπάρχουν πολλές δυνατότητες και καλά παραδείγματα στα οποία μπορούν να ε, επέμβουν οι τοπικές αρχές ε, που εν τέλει θα εκμεταλλευτούν την προστιθέμενη αξία την οποία θα έχει κερδίσει το ανανεωμένο, ανακαινισμένο οίκημα. και ε, βεβαίως ε, για την ε, νεολαία, για τους νέους, νομίζω ότι, όπως είπε και ο κύριος Πετριτσόνε, γιατί να μην ζητήσουμε από το Κοινοβούλιο να διοργανώσει ε, ένα μεγάλο διάλογο με τη νεολαία, ε, γιατί οι νέοι διαδηλώνουν, κάνουν αυτές τις πορείες, τις διαδηλώσεις για το κλίμα ε, και επομένως ε, βλέπουμε πλέον ότι οι άνθρωποι ξέρουν πού θέλουν να πάνε, με ποιο τρόπο, ποιες είναι οι ιδέες τους, είναι συγκεκριμένες. Επομένως, ε, να ε, πιέσουμε έτσι ώστε να υπάρξει ένας διάλογος υψηλού επίπεδου. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ όλους τους παρεμβαίνοντες. Αποχαιρετούμε τους συμμετέχοντες στο πάνελ και γιατί πρέπει να συνεχίσουμε και με τις συνήθεις εργασίες μας. <clears throat> Ε, προχωράμε με την επόμενη έκθεση που είναι η ε, μακροπρόθεσμη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά ε, τα, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Δίνω πρώτα το λόγο στον κύριο Πίτερ Λίζε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρόκειται πλέον για το συγκεκριμένο κείμενο το οποίο θα ψηφίσουμε στην ε, Επιτροπή μας. Εγώ προσωπικά δηλώνω ικανοποιημένο από την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, διότι το βασικό αίτημα του ψηφίσματος και το βασικό αίτημα του ψηφίσματος μάλλον, το οποίο έχω υπογράψει, συζητούμε μέσα στην ομάδα μου του Λαϊκού Κόμματος και θα πρέπει να συνεργαστούμε και με άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπέ, ώστε όταν φτάσουμε και στην Ολομέλεια να το κάνουμε αυτό και πιο εντατικά. Ακόμα δεν υπάρχει ορατή τελική ε, ε, εκδοχή ας πούμε. Αν είναι να φτάσουμε στην Ολομέλεια πρέπει να εμπλακούν και άλλες άλλε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ. Αυτό που με εντυπωσιάζει στο έγγραφο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το είπα και στην ακρόαση είναι ότι η Επιτροπή λέει ότι μπορούμε να αναμένουμε κέρδος, καθαρό κέρδο ενό εκατομμυρίου θέσεων εργασία. Αυτή τουλάχιστον η στρατηγική δεν θα οδηγήσει σε απώλειε απασχόληση. Τώρα, εάν είναι ένα εκατομμύριο ή παραπάνω θέσει εργασία ή 500.000 ή και λίγο παραπάνω από ένα εκατομμύριο, αυτό μπορεί ίσω να ε, το υπολογίσει κανεί με διαφορετικού τρόπου. Αλλά πρόκειται για μια σαφέστατη και ε, σημαντική δήλωση, την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν την κάνει χωρί βάση. Είναι σημαντικό λοιπόν να λεχθεί. Για μα, ω Λαϊκό Κόμμα, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είναι σημαντικό η παραγωγή χωρί εκπομπές διοξιδίων του άνθρακος, παραγωγή ε, προϊόντων ε, εντάσσεως ενέργειας, είναι πολύ σημαντική υπόθεση και η δίκαιη μετάβαση, just transition, transition, την οποία έχουμε περιλάβει στο σχέδιο του ψηφίσματος, αλλά νομίζω πρέπει να το ε, διατυπώσουμε με ακριβέστερο τρόπο. Έως τώρα, από Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Συμβουλίο, ακούμε μεν ωραία λόγια, δεν βλέπουμε όμως συγκεκριμένα, συγκεκριμένους πόρους να διατίθεται. Γι' αυτό και θέλουμε να πούμε συγκεκριμένα εμεί ότι στο ΠΔΠ θέλουμε να δούμε κονδύλια δεσμευμένα ειδικά για τους σκόπους αυτούς. Όχι μετά από 15 αιτήσει. Πρέπει να είναι σαφές ότι τα χρήματα αυτά προβλέπονται να διατεθούν για την δίκαιη μετάβαση. Για μένα το πιο σημαντικό, το απολύτω πιο σημαντικό είναι να καταλήξουμε σε ευρύτατη πλειοψηφία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τον τρόπο αυτό να παρακινήσουμε και το Συμβούλιο στην διάσκεψη κορυφή του Σίβιου, να υποστηρίξετε τη γη αυτή και να προετοιμάσετε τα επόμενα βήματα. Το Σίβιου θα τεθεί ως θέμα το μέλλον της Ευρώπης. Δεν είναι δυνατόν εκεί η προστασία του κλίματος να μην διατυπωθεί σαφώς μέσα στην δήλωση που θα προκύψει από τις εργασίες του Σίβιου. Επειδή λοιπόν είναι τόσο σημαντικό το θέμα, παρακαλώ οι συνάδελφοι να σκεφτούν πραγματικά αν όντως θέλουν να βάλουν και χίλια άλλα πράγματα μέσα στο ψήφισμα αυτό ή αν μπορούμε ίσως να τα συζητήσουμε ήσυχα μετά τις ευρωεκλογέ. Επομένως, 55% για το 2030, το 45% για το 2030 τα έχει αποφασίσει το Συμβούλιο και με σύμφωνο, και το Κοινοβούλιο, συγγνώμη, με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αλλά θα αποτρέψει πολλές χώρες αν βγούμε τώρα να μιλήσουμε για 55% προτείνω ε, να ε, ασχοληθούμε περισσότερο με την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, ίσως μπορούμε να υπερβούμε και το 40% χωρίς να το παρακάνουμε. Νομίζω επίσης ότι δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή, στο παρόν ψήφισμα δηλαδή, να συζητήσουμε για το τι θα γίνει στο, στην αναθεώρηση 2022-2023 υπήρξαν προτάσεις από συναδέλφους σχετικά με την ενίσχυση των στόχων για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος από ε, επιβατικά αυτοκίνητα. Αλλά αυτό νομίζω πρέπει να το συζητήσουμε περισσότερο πριν να το ε, βάλουμε στο ψήφισμα. Και υπήρξαν και προτάσεις να μιλήσουμε για, για 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2050. Και αυτό νομίζω ότι είναι πρόημο. Άλλωστε είναι και αρμοδιότητα της Επιτροπής Ήτρε. Να είμαστε λοιπόν λίγο πιο αυτοσυγκρατημένοι. Τελευταίο, για να αποδώσουν όλα αυτά και ιδίω για να σταθεροποιηθεί το κλίμα και να επιτευχθούν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι θερμοκρασίας του Παρισιού, πρέπει να ενισχύσουμε την διεθνή διάσταση. Στην Ευρώπη διεξάγεται συζήτηση για τους στόχους 2050 με συγκεκριμένα μέτρα που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένες στρατηγικές. Διεξάγεται εδώ λοιπόν μια συζήτηση και πολύ εντατικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προσαρμογή των στόχων 2030 που όμως σε, στις άλλες μεγάλες οικονομίες δεν βλέπουν να διεξάγει τέτοια συζήτηση έθεσα συστηματικά το ερώτημα στη διάσκεψη του κλίματος για τη Βόνια αλλά και στην Κάτοβιτς. Πού έχετε φτάσει σε ό,τι αφορά τους στόχους 2030. Με κοιτούσαν κατάπληκτοι. Δεν γνώριζαν καν περί τίνο ομιλούσα. Αυτοί θεωρούν ότι αρκεί να ικανοποιήσουν τους στόχους της Συμφωνία του Παρισιού και ούτω ή άλλως αυτούς δυσκολεύουν αρκετά. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε να μην δώσουμε την εντύπωση στον κόσμο ότι αν η Ευρώπη επιτύχει τους στόχους που έχει βάλει, έχει σώσει το κλίμα. Χρειάζονται πολλέ σχέσει και με τι άλλε χώρε και δεν μιλώ βεβαίω μόνο για τη Βραζιλία και τι ΗΠΑ, όπου εκεί υπάρχει σαφέστατη η παναχώρηση από του στόχου, αλλά και για Ιαπωνία, Μεξικό και άλλε μεγάλε οικονομίε. Πρέπει να ρίξουν περισσότερο βάρο εκεί λοιπόν. Ευχαριστώ. Έχει τώρα το λόγο η κυρία Γκούτελάντα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε η οι δημοκράτες, οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες ε, βλέπουν με πολύ θετικό βλέμμα την πρόταση της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει πολύ συγκεκριμένους στόχους και όντως μέχρι το 2030 να επιτύχει αυτήν την ουδετερότητα. Οπωσδήποτε χρειαζόμαστε βιώσιμο μέλλον και για την Ευρώπη και για τον υπόλοιπο κόσμο και θα πρέπει για να το επιτύχουμε να εφαρμόσουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους βιώσιμης ε, ανάπτυξης. Το κόστος της μη ανάληψης ε, δράσης είναι πολύ βαρύ. Είναι απαράδεκτο ε, για να βαρύνουμε με αυτήν την μη απόφαση την ανθρωπότητα. Το θέμα δεν είναι μόνο να έχουμε λιγότερες εκπομπές, αλλά αυτό να γίνει με έναν δίκαιο τρόπο. Τρία είναι τα κύρια στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, ο, το κλίμα θα πρέπει να λειτουργήσει σε μία ε, ε, κοινωνία που ιδεολογικά και κοινωνικά θα είναι βιώσιμη. Ε, όλοι μαζί δηλαδή θα πρέπει να φτάσουμε στον στόχο αυτό. Εμείς βλέπουμε και μεγάλες ευκαιρίες για την Ευρώπη. Συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λέει ότι θα προκύψουν μεγάλες ευκαιρίες για την απασχόληση. Αλλά θα πρέπει ε, θα πρέπει να ε, ανακυκλωθούν εργασιακά και όλοι αυτοί οι οποίοι θα βρεθούν χωρίς απασχόληση λόγω των τεχνολογιών κλπ. Θα πρέπει οπωσδήποτε λοιπόν με δίκαιο τρόπο να γίνει αυτή ε, η αλλαγή. Ο κύριος Λίζε είπε πολλά σωστά πράγματα, αλλά η περισσότερη δουλειά όσον αφορά αυτά τα ωραία λόγια ακόμα δεν έχει γίνει. Τον Μάιο το Συμβούλιο κατέδειξε ότι η θέση του Κοινοβουλίου είναι πολύ συγκεκριμένη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προχωρήσει και να προοδεύσει η Ευρώπη. Ε, μέχρι το 2050 θα πρέπει να έχει ξεκαθαριστεί το τοπίο και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η μετάβαση. Είναι τελικά πολύ πιο ακριβό πλέον, κοστίζει πολύ περισσότερο να έχουμε μια οικονομία με τέτοιες εκπομπές παρά μια οικονομία χωρίς. Εμείς ε, θα υποβάλουμε ως σοσιαλιστές και δημοκράτες κάποιες τροπολογίες ε, έτσι ώστε ε, να μειωθούν με ταχύτερο ρυθμό οι εκπομπές. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει οι στόχοι να είναι πιο αυστηροί και οπωσδήποτε να ευθυγραμμίζονται με τους ιδιαίτερα μακροστρο... μακροπρόθεσμους στόχους και οπωσδήποτε θα πρέπει να συμβάλλει και η βιομηχανία σε αυτήν την τροποποίηση και σε αυτήν την μετάβαση. Ε, δεύτερον, ε, οι βιομηχανίες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα μείωσης πιο γρήγορα θα πρέπει να το κάνουν. Επίσης στις ε, οικοδομές ε, θα πρέπει να προωθηθούν οι λύσεις αυτές οι οποίες είναι πιο αποδοτικές ε, ενεργειακά. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν ολόκληροι τομείς οι οποίοι να μην κάνουν καμία προσπάθεια. Ούτε είναι σωστό ένας και μόνο τομέας να επομιστεί όλη την προσπάθεια. Θα πρέπει να ενδυναμώσουμε επίσης τη δασοπονία γιατί ξέρουμε ότι τα δέντρα έχουν την ικανότητα να απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακος και να αποδίδουν στην ατμόσφαιρα οξυγόνο. Θα πρέπει οπωσδήποτε να μειωθεί, να απαλληφθεί η χρήση των ε, ορυκτών καυσίμων. Όλα αυτά όμως θα πρέπει να γίνουν όπως ε, είπα και προηγουμένως με δίκαιο τρόπο, δίκαιο για όλους ε, και γι' αυτό είναι καλό να υπάρχει ειδικό ταμείο για ε, κοινωνικώς αποδεκτή ε, κλιματική μετάβαση. Οι δε περιφέρειες οι οποίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα ε, μεγάλες προκλήσεις θα πρέπει να βοηθηθούν. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε καλές και προοδευτικές λύσεις για την Ευρώπη και το κλίμα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος θα περάσω αμέσως στον κύριο Έικχουτ, γιατί οι δύο επόμενοι σκιώδεις λείπουν. Thank uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω οι δύο συναδελφοί μου, οι προαλήσαντες, εξήγησαν τη σημασία του όλου θέματος και εγώ θα ήθελα να προσθέσω σε όλα αυτά ότι δεν πρόκειται μόνο για την 9η Μαΐου, όπου ε, οι αρχοί κρατών και θα μιλήσουν για το μέλλον της Ευρώπης. Βεβαίως και το μέλλον της οικονομίας μας ε, είναι καθοριστικό θέμα. Στις 23 Σεπτεμβρίου του 19 μετά θα ακολουθήσει δεύτερη συνάντηση όπου ε, ο κόσμος περιμένει κάτι, από όλο τον κόσμο περιμένει κάτι και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πάμε στη Νέα Υόρκη και τώρα που προετοιμάζουμε το ψήφισμα είναι κατάλληλη στιγμή να πούμε κάτι από αυτού. Εφόσον χαράσουμε μακροχρόνια στρατηγική, βεβαίως και αυτό θα επηρεάσει το τι υποσχόμεθα σε ολόκληρο τον κόσμο. Και μπορώ και να σας παραθέσω το τι είπε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών που λέει ότι επιθυμούμε οι χώρες να είναι λίγο πιο φιλόδοξος στην κλιματική αλλαγή. Τέλος της παράθεσης. Ε, στις 23 Σεπτεμβρίου ο κύριος Γκουτιέρες θα ε, συνενώσει τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Ε, οι άνθρωποι θα παρακολουθούν το τι θα κάνει η Ευρώπη και αν απλά έχουμε μια γενική συζήτηση για μακροχρόνια στρατηγική όπου δεν υπάρχει καν αυτή η συζήτηση γιατί το έγγραφο της Κομισιόν είναι μία ανακοίνωση που ανοίγει τη συζήτηση για τη μακροχρόνια στρατηγική. Άρα δηλαδή αυτό δεν είναι στρατηγική, είναι η έναρξη. Αρχίζει η συζήτηση για το πότε θα ακολουθήσει η στρατηγική. Και αυτή είναι η γραμμή μας ως Ευρώπη ε, για το Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη. Αυτό πολύ λίγο ελάχιστο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Πίτερ, θέλω να σου πω ότι ήσουν σε άλλο Κατοβίτσε αυτό που, αυτό που ήμουν εγώ, γιατί στο Κατοβίτσε ε, συνεχώς γιατί το θέμα για το τι μπορούμε να κάνουμε ε, για να βελτιώσουμε τους αναπτυξιακούς στόχους. Ίσως να μην τα άκουσες αυτά. Πάντως, ε, ε, στα Ηνωμένα Έθνη όλες οι χώρες είναι ίδιες. Το να λέει κανείς <laughs> αυτή είναι μικρή χώρα ε, και δεν μετράει γνώμη της, εντάξει, την προσβάλλεται κιόλας. Εάν μια μεγάλη οικονομία όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προχωρήσει, τότε μπορούμε ήδη τώρα να συμπεράνουμε ότι όχι μόνο ο Σεπτέμβρης θα αποτύχει, αλλά προτιμάζουμε την αποτυχία και για αργότερα. Δεν είναι λοιπόν κατάλληλη στιγμή για να είμαστε αυτάρεσκοι. Υπάρχουν ορισμένα θέματα ε, σε μια πολιτική ομάδα γιατί δεν μπορούν να καταλήξουν σε νέα θέση. Αλλά ξέρετε, σε τελική ανάλυση αυτό που διακυβεύεται είναι το τι χρειαζόμαστε για το κλίμα να ακολουθήσει ε, μια ε, βελτίωση αν θέλουμε να παραμείνουμε μέσα στους στόχους μας. Μείωση κατά 1,5 Άρα δηλαδή να είμαστε πιο φιλόδοξοι, η μακροχρόνια στρατηγική βοηθάει, αλλά είναι άχρηστη αν όλα αυτά δεν τα μεταφράσουμε σε πράξεις. Και οι άνθρωποι ζητάνε απαντήσεις τώρα. Παντού διαβάζω ότι οι μαθητές ε, εξεγείρονται, αλλά δεν λένε ότι θέλω στρατηγική για το 2050, δεν το διάβασα ποτέ αυτό. Τώρα λέει, τώρα θέλω. Και ήρθε η ώρα οι πολιτικοί να τα ακούσουν αυτά και μέσα σε ψήφισμα να βάλουν ιδέες για το μέλλον. Εμείς ως Κοινοβούλιο το έχουμε ήδη κάνει και θα ήταν πολύ δυσάρεστο ως Κοινοβούλιο να υπαναχωρήσουμε σε κάτι επί το οποίο συμφωνήσαμε το Δεκέμβρη. Ε, συγγνώμη Πίτερ, αλλά θα γίνει συζήτηση και υπάρχει ευκαιρία ε, για το ΕΛΚ να συμμετέχει και αυτό. Αλλιώς θα είσαστε από εκείνου ε, ε, που δεν θέλουν τίποτα. Δεν ξέρω το αν σας αρέσει να στριμωχτείτε σε αυτή τη γωνία. Άρα δηλαδή είναι ανοιχτή η πρόσκληση να έρθετε μαζί μας και η Ευρώπη να γίνει πιο ελκυστική καθώς θα πηγαίνουμε στη Νέα Υόρκη και όχι να γίνει ενοχλητική. Αυτό πρέπει να το απαντήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Τελευταία θα πάρει το λόγο η κυρία Ελεονόρα Εύη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερος. Τι να πω. Σύμφωνα με την έκθεση της IPCC, που ήταν σαφέστατο, ε, είναι συγκεκριμένο ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας έτσι ώστε να βρούμε λύση. 12 χρόνια είναι ο χρήσιμο χρόνος για να φτάσουμε στο σημείο χωρίς επιστροφή. Ε, όπου οι καταστροφές δεν θα έχουν πραγματικά δυνατότητα αντιστροφής. Ε, και ο Ζανσο Φωσάικουτ τα είπε προηγουμένως και άλλοι συνάδελφοι. Εδώ έχουμε ένα ψήφισμα το οποίο θα πρέπει να θέσει τις βάσεις ε, για την συζήτηση που δεν μπορεί να παραμείνει μόνο συζήτηση αλλά θα πρέπει να υλοποιηθεί μέσα από συγκεκριμένε δράσεις. Η Ευρώπη θα πρέπει να αποφασίσει ποιο δρόμο θέλει να πάρει και στα διεθνή φόρα να το πει με ε, ε, πολύ σαφή, σαφή τρόπο. Αλλά με την ίδια σαφήνεια θα πρέπει να το τονίσει και στα ενδοευρωπαϊκά φόρα. Δεν πρέπει να φοβόμαστε ε, να έχουμε φιλόδοξες θέσεις Έχουμε πληθώρα ε, ε, νομοθετικών εγγράφων, κανονισμών, οδηγιών ε, και για τις μεταφορές και για άλλα. Και εδώ επαναλαμβάνουμε και ξαναλέμε ότι είναι πολλοί αυτοί οι τομείς οι οποίοι τα τελευταία χρόνια με γεωμετρική πρόοδο έχουν αυξήσει την εκπομπή αερίων και επομένως εκεί χρειάζεται αντιμετώπιση με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα έτσι ώστε να έχουμε μεγάλη μείωση ε, και να μειωθούν, ε, να συμμικρωθούν και τα κόστη ε, στους τριμερείς διαλόγους, στις εργασίες, στο Συμβούλιο βεβαίως. Δεν καταλαβαίνουμε πολύ καλά πώς λειτουργούν τα πράγματα ή μάλλον αντιθέτως τα καταλαβαίνουμε πολύ καλά και ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να κατεβάσουν το επίπεδο των φιλοδοξιών. Ε, ο τομέας ε, των μεταφορών λοιπόν είναι μεταξύ αυτών των τομέων που θα πρέπει ε, να διευθετείται από πιο αυστηρούς φιλόδοξους κανόνες. Είναι απαραίτητο, όπως αναφέρεται και στο ψήφισμα που εκπονήσαμε, είναι απαραίτητο, λέω, να υπενθυμίσουμε τους ε, μέσο πρόθεσμους στόχους ε, και οπωσδήποτε αυτός ο στόχος να είναι όσο γίνεται πιο ευθυγραμμισμένος με τους μακροχρόνιους ε, στόχους. Επίσης, η έννοια της δίκαιης μετάβασης επιτέλους αρχίζει και σηκώνει κεφάλι. Ε, πρώτα για τα αυτοκίνητα ας πούμε που ε, ίσως για μία φορά επιτέλους υπογραμμίζεται η ανάγκη ε, της κάλυψης της απασχόλησης και των κοινωνικών αλλαγών. Εδώ οδηγούμεθα λοιπόν στην αναγνώριση ότι θα πρέπει να αλλάξει το υπόδειγμα θα πρέπει οπωσδήποτε να εγκαταληφθούν κατά προτεραιότητα ή ε, τα ορυκτά καύσιμα και κάτι άλλο ε, που πρέπει οπωσδήποτε κατά την άποψή μου στο ψήφισμα αυτό να βρει τη θέση του. Είναι το εξής, ε, ποιο δρόμο θέλουμε να ακολουθήσουμε μετά το 2030 με για το, μετά το 2030 για το ETS, αυτό το σύστημα το οποίο ε, ξεκίνησε από την Ευρώπη και πλέον έχει διαχειριστεί σε ολόκληρο τον κόσμο και που δεν μπορεί να αποτελέσει τη μοναδική οδό Ε, δεν είναι πολύ αποτελεσματικός, ε, ε, αποτελεσματικός τρόπος για να μειωθούν οι εκπομπές. Από τη μία μεριά θα πρέπει να μειωθούν πραγματικά οι εκπομπές και μετά θα πρέπει να αξιολογήσουμε την παραγωγή που γίνεται εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που είναι οπωσδήποτε πιο καθαρή από την παραγωγή αλλού. Τέλος, τέλος και πραγματικά τελειώνω με αυτό. Η, γεωργία δεν είναι δυνατόν να είναι πάντα απούσα. Έχει το μεθάνιο, έχει μια σωρό, ένα σωρό ε, ουσίες ε, τις ε, οποίες εκλείει ε, και επομένως δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε συγκεκριμένους και σαφείς κανόνες και όσον αφορά το θέμα αυτό. Ωραία, μίλησαν λοιπόν οι συνεισηγητές, ε, δεν έχει ζητήσει κάποιος ε, το λόγο, από ό,τι, από καταλαβαίνω δεν θέλει κάποιος να μιλήσει. Ε, γι' αυτό λοιπόν σας λέγω ότι 31 ε, Ιανουαρίου, 5 το απόγευμα, προθεσμία υποβολής τροπολογιών, μόνο στα αγγλικά. Ε, ψηφοφορία στην Έμβη 20 Φεβρουαρίου του 19 και ψηφοφορία στην Ολομέλεια τον Μάρτιο στην πρώτη ή στη δεύτερη ολομέλεια του Μαρτίου. Α, τη δεύτερη ολομέλεια του Μαρτίου μου λέει η γραμματεία. Σας λέγω επίσης ότι οι επόμενες συνεδριάσεις θα λάβουν χώρα την 7η Φεβρουαρίου 2019 στις 9. Θα έχουμε κοινή με την ΕΝΤΕΒΕ δημόσια ακρόαση όσον αφορά τους στόχους ε, βιώσιμης ανάπτυξης 2018. Δεν έχουμε ακόμα την ακριβή αίθουσα. Επίσης, κοινή NVDEV, συνεδρίαση επιτροπής, ε, σύμφωνα με τον κανόνα 52, όσον αφορά ε, την υλοποίηση των ε, ετήσιων στόχων, όσον αφορά, συγγνώμη, την ετήσια έκθεση για την υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτά και τελείωσε η συνεδρία σήμερα.